Καλησπέρα, συνάδελφοι. Ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Ας προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Πάρτε θέσει για να ξεκινήσουμε, να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, καθίστε και με ησυχία. Δεν είναι ακόμα πλήρη η αίθουσα, είναι προφανές, αλλά ξέρετε πώς είναι τα πράγματα, είναι ολομέλεια. Ταυτόχρονα έχουμε και αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Οπότε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Έχουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα επικεντρωθεί στην ακρόαση τριών υποψηφίων που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Επιλογής για τη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Πρώτα λοιπόν πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ποια είναι η γλωσσική κατάσταση στην ε, συνεδρίασή μας. Όλες οι γλώσσες εκτός από ε, κροατικά, ε, αλικιανά, λιθουανικά και μαλτέζικα. Σύμφωνα τώρα με τα όσα λάβαμε από, ως σημειώσεις από την συνεδρίαση των συντονιστών, ε, υπάρχουν κάποια, κάποιες συστάσεις ε, τις οποίες ε, θα ήθελα να εγκρίνουμε. Κύριε Πουσαδευλίκα, είδα το χέρι σας. Για το 2.14 του κανονισμού και σχετικά με την απόφαση των συντονιστών, να μην συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε σχέση με τη συμπερίληψη κάποιων ομάδων στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Θα ήθελα να ζητήσουμε από το Συμβούλιο τη συμπερίληψη μιας συγκεκριμένης οργάνωσης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε στο Συμβούλιο την προηγούμενη συνάντηση. είναι κάτι το είναι πάρα πολύ γνωστό. Υπάρχουν έτσι και αλλιώ ε, επτά ε, υποκράτηση μέλη της συγκεκριμένη οργάνωσης για επιθέσεις εναντίον ε, των πολιτικών και έχουν βρεθεί και σχέδια για απειλές ενεργειών εις βάρος ε, της Ισπανίας, ε, της Γαλλίας, ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας στα πλαίσια του Σέγγεν, λιμένων, αερολιμένων κτλ. Είναι μια απειλή για τη δημοκρατία και καλό θα είναι να μπορέσουμε να συζητήσουμε και τα θέματα τα οποία ανήκουν στις αρμοδιότητες μας. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουσαρέρα, αλλά σας θυμίζω ότι το 2014 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέει ότι οι συντονιστές είναι αυτοί οι οποίοι στις τακτικές συνεδριάσεις τους οι οποίοι θα αποφασίσουν για τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου ε, θέματος στην ημερήσια διάταξη και ε, η πλειοψηφία των συντονιστών αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσείς θέλετε να ψηφίσουμε γύρω από την απόφαση των συντονιστών και αυτό το οποίο εγώ προτείνω είναι η ψηφοφορία αυτή να γίνει αύριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι αύριο στις 10 το πρωί θα πρέπει να είμαστε παρόντες εδώ με τις ηλεκτρονικές μας κάρτες για να ψηφίσουμε επί των υποψηφίων οι οποίοι σήμερα θα περάσουν από ακρόαση από την Επιτροπή μας. και θα ξεκινήσουμε επίσης ε, με την υπεύθυνη ε, προτινόμενη για την υπηρεσία προστασίας της ιδιωτικότητας. Πράγματι ε, βλέπω τώρα ότι αυτό έχει συμπεριληφθεί στην αυριανή συνεδρίαση αλλά λόγω της σημασίας που έχει το θέμα και επειδή έχουν περάσει τρεις συνεδριάσεις που δεν συζητήσαμε το θέμα αυτό, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι για να υπάρχει διαπαρτία σε σχέση με την συζήτηση. Για να διευκολύνω ακριβώς το δικαίωμα ψήφου όλων των μελών, έχουμε ανακοινώσει ότι αύριο στις 10 το πρωί με τις ηλεκτρονικές κάρτες θα μπορέσουν τα μέλη να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία κάτω από τις σωστές συνθήκες. Το θέμα είναι ότι εμείς εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών, όπως έγιναν δεκτές, τις συστάσεις τους, ε, αλλά ε, το θέμα εδώ είναι μια πρόταση του ECR και η πρόταση αυτή θα ψηφιστεί αύριο από το σύνολο των μελών, αύριο το πρωί στις 10. Κατά τα άλλα, οι προτάσεις των συντονιστών δεν την χάνουν αντιρρήσεων και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε. Όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Έχουμε ένα θέμα λοιπόν στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση. Να προχωρήσουμε στην ακρόαση των υποψηφίων ε, για την θέση της Υπηρεσίας Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε τι λέει ο κανονισμός από το 18. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο διορίζουν τον υπεύθυνο, το EDPS θα το λέμε από εδώ και πέρα, μετά από συνένεση, μετά από κοινή γνώμη. Αυτό σημαίνει ότι καταρχάς το Συμβούλιο ψηφίζει ε, ε απόρριτα, Έγινε η ψηφοφορία την προηγούμενη εβδομάδα και γι' αυτό μένει εμείς πλέον να κάνουμε ε, την δουλειά που μας αναλογεί. Θα ακούσουμε 45 ε, λεπτά τον καθένα τους τρεις ε, υποψηφίους που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <coughs> Έχω εδώ τα τρία ονόματα. Και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω ε, κάποια ή κάποια συνάδελφο να βγάλει το πρώτο όνομα το οποίο θα ακούσουμε και μετά οι υπόλοιποι δύο θα ακολουθήσουν με αλφαβητική σειρά. Ο πρώτος όμως ο οποίος θα πάρει το λόγο είναι ο η, Τσάμπο, Έντερτ και μετά θα ακούσουμε τους άλλους δύο υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Πάντοβα δηλαδή ο δεύτερος. Yes. Yes, but this is the first one. This is the first one, is it not? Yes. And then the second one will be? Συγγνώμη, η αλφαβητική σειρά καθορίζεται από τον πρώτο ε, που επελέγει. Ζάμπο ο πρώτος, Βεβερόφσκι ο δεύτερος και Πάντοβα ο τρίτος. 45 λεπτά μέγιστος χρόνος για τον κάθε έναν από αυτούς. 5 λεπτά για μια σύντομη παρουσίαση των απόψεών τους για την υπηρεσία και μετά ερωταπαντήσεις Δέκα ερωτήσεις, ε, μέγιστος αριθμός. Ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε δίκαια και σύντομα τον χρόνο. 45 λεπτά για τον καθένα. Έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν. Να σας υπενθυμίσω ότι η εντολή της ηγεσία του EDPS τερματίζεται στις 5 Δεκεμβρίου. Πάρα πολύ σύντομα λοιπόν. Ξεκίνησε τον Απρίλιο στις 11 Απριλίου η διαδικασία κάλυψης της θέσης, η προθεσμία ήταν 16 Μαΐου, αλλά ο σύντομος κατάλογος των επιτυχόντων μας απεστάλλει στις 30 Οκτωβρίου, δίδοντάς μας ελάχιστο χρόνο έτσι ώστε να αξιολογήσουμε τους υποψηφίους και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέχρι κοινή μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό λοιπόν συνεδριάζουμε εκτάκτος σήμερα και γι' αυτό θα ψηφίσουμε αύριο εκτάκτος πάλι <clears throat> στις 10 το πρωί. Παρακαλώ πάρτε τις κάρτες σας όλοι αύριο μαζί. And I, I, uh, uh, understand... Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένας κατάλογος ονομάτων που έχουν ήδη καταχωρηθεί για την υποβολή των ερωτήσεων. Ο καθένας έχει ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο, λεπτά για την απάντηση, δέκα ερωτήσεις συνολικά στη σειρά και μέγιστο αριθμός δέκα. Έχω τον κατάλογο. Από ό,τι βλέπω έχουν συμφωνήσει οι συντονιστές να ανατεθεί ο χρόνος ε, των ερωτήσεων για να είναι, είμαστε δίκαιοι για όλους, για να ακούσουμε στον ίδιο χρόνο από όλους τους υποψήφιους. Ο κύριος Ζάμπο είναι καθοδόν από ότι με πληροφορούν. And, uh, Όπως ε, γνωρίζουμε όλοι. Ε, αυτή τη στιγμή ε, έχει ξεκινήσει η όλη ομέλεια και πραγματικά θα εκτιμούσα τη συνεργασία σας να χειριστούμε ομαλά και δίκαια αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να είμαστε δίκαιοι με όλους. Ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση για να ε, χειριστούμε όλους τους υποψήφιου με ίσο τρόπο. Κύριε Ζάπο, καλώς ορίσατε. Please be welcome. have you here. Thank you very much.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 Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλωσορίζουμε θερμά τον κύριο Ζάπο. Έχετε επιλεγεί με κλήρο ως πρώτος υποψήφιος, τον οποίο θα ακούσουμε εδώ. Λοιπόν, ε, τραβήξαμε κλήρο από το φάκελο αυτό και τώρα είναι η σειρά σας να κάνετε μια δήλωση, όχι πέραν των 5 λεπτών. Μετά 10 μέλη θα σας υποβάλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις διάρκειας ενός λεπτού και θα έχετε δύο λεπτά να απαντήσετε σε κάθε μία ερώτηση. Συνολικά 45 λεπτά. 45 λεπτά και οι τρεις υποψήφοι. Σας συγχαίρω λοιπόν που ε, έχετε επιλεγεί από την Επιτροπή Επιλογής, διότι πιστεύω ότι είναι μια επιτυχία από μόνη της. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, λοιπόν. Thank you very Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ που με κληρώσετε πρώτο. Ε, έχετε τυχερό χέρι και το θεωρώ θετικό ιονό. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σα εδώ για ε, να ε, παρουσιαστώ ενώπιον τη Επιτροπή. Όπω ξέρετε, ω υποψήφιο είχα μια σειρά από συναντήσει πρωτού παρευρεθώ εδώ και τόνισα στην επιστολή μου ότι έχω προσιλωθεί στο να εξυπηρετήσω του πολίτε για, για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Και έχω τώρα την ευκαιρία να συναντηθώ κατευθείαν με τους εκπροσώπους που εκλέγονται κατευθείαν από τους πολίτες. Απέναντί σας έχω την ευκαιρία ε, να αντιμετωπίσω ε, κατά μέτωπο τους ίδιους τους πολίτες του οποίους θα εξυπηρετήσω. Άρα για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική από όλες ε, τις συναντήσεις που είχα μέχρι στιγμής. Και μιλάω με ευθύνη και δέσμευση προς Όπως είδατε στο βιογραφικό μου, η σταδιοδρομία μου έχει σχέση στενή με θέματα προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη. Δούλευα ως ε, Εθνικός Εμπειρογνώμονας ε, στο EDPS το 2006 και 2007. Μετά από μερικά χρόνια ήμουν επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την προστασία των ε, δεδομένων στο Συμβούλιο και τότε είχα μια, συνομιλία με κάποιον από εσά σε αυτή την Επιτροπή. Ως ε, ε, πρόεδρος ήθελα να ακούσω την προοπτική του Ευρωκοινοβουλίου και ήμουνα πάντοτε καλός στο να ακούω τους άλλους. Και το τρίτο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ο ρόλος μου Εντό του Συμβουλίου Προστασία των Δεδομένων. Ήμουν κεφαλή της ε, υπομάδας ε, των εμπειρογνωμόνων με την εμπειρία ε, που έχω είμαι σε καλή θέση να έχω την θέση του επόμενου Ευρωπαίου Επόπτη Προστασία Δεδομένων. Οι επιτυχίες μας στον τομέα της ιδιωτικής ζωής είναι ένα μέρος τη μεγαλύτερη εικόνα. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που έχουμε πετύχει. Έχουμε το πιο δυνατό και φιλόδοξο πλαίσιο προστασίας δεδομένων στον κόσμο. Παρόλο που ακόμη λείπουν ίσω κάποια δομικά στοιχεία. Αναμενόμαστε να ε, προστατεύσουμε αυτό το κομμάτι του κεκτημένου προς όλους, προς τρίτους και προς συμμετόχους στο τομέα των επιχειρήσεων. Η ιδιωτικότητα των προϊόντων μας δεν μπορεί ποτέ να, ε, είναι θέμα συμβιβασμού. Και γνωρίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας εταίρος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ε, οι δραστηριότητες σα σε αυτό τον τομέα είναι εντυπωσιακέ. Ε, οι αρχές εποπτείας προστασίας των δεδομένων είναι πολύ δραστήριες σε αυτό τον τομέα. Η θητεία μας και η εντολή μας θα είναι ε, πάντα απέναντι στους πολίτες και έχουμε πάντα την υποψία ότι το μολυστικό παιχνίδι που παίζουν κάποιοι γίγαντες της τεχνολογίας είναι προς, ε, ε, εις βάρος των πολιτών. Ο ανταγωνισμός και η ιδιωτική ζωή εδώ ε, συναντιόνται, αλλά η προστασία των δεδομένων των πολιτών ε, πάνε πολύ περισσότερο από τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Όπως έχει δείξει και το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, διακυβεύονται οι κοινωνίες μας. Πάντα προχωρούμε ε, αν αναλαμβάνεται περισσότερος έλεγχος των δεδομένων και τώρα πρέπει να κρατούμε τα μάτια μας ανοιχτά όχι μόνο στις κυβερνήσεις αλλά και σε άλλους ε, παίκτες, ιδιαίτερα αυτούς για τους οποίους η ιδιωτικότητα έχει διαφορετική αξία από ό,τι κατανοούμε εμείς. Ο ρόλος ε, του επόπτη και των αρχών προστασίας ε, δεδομένων συμπεριλαμβανομένου του EDPS ε, χτίζεται σε μια κουλτούρα προστασίας των δεδομένων και δεν πρέπει να υποεκτιμάται. Ο EDPS αμφίβολα συγχωρεί υπέρ της προστασίας των δεδομένων των πολιτών της Ευρώπης δεν είναι δική μου φιλοδοξία ως υποψήφιο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Όταν ε, υπέβαλα την υποψηφιότητά μου, ε, έλαβα υπόψη μου και αυτό το μελλοντικό μου ρόλο. Κυρίε και κύριοι, είμαι έτοιμο να δουλέψω μαζί σα για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία τη ιδιωτικότητα για την ευημερία των πολιτών μα. Προσβλέπω στις ερωτήσει σα και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Κύριε Πρόεδρε, εδώ κλείνει η εισαγωγή μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσατε στον στο χρόνο σας. Τώρα ας προχωρήσουμε. Χρόνος ερωτήσεων. Ξεκινούμε με την κυρία Μετσόλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή, ενώ το θεσμικό και νομικό πρόβλημα, ε, πλαίσιο ε, υπάρχει. Υπάρχουν και οι κανόνες για την αμοιβαία συνδρομή από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Οι ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικές αρχές σε διασυνοριακές καταστάσεις είναι μεγάλες. Ε, βάσει αυτού του κανονισμού που μόλις ανέφερα, ο επόπτης θα πρέπει να συνεργάζεται με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Βλέπετε κάποια περιθώρια βελτίωσης στην αντιμετώπιση αυτού του ρόλου και αν εσείς επιλεγείτε πώς ε, θα διασφαλίσετε ότι οι διάφορες αρχές προστασίας δεδομένων θα έχουν μια συνεκτική προσέγγιση στην ερμηνεία και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αλλά θα γίνεται σεβαστή και ανεξαρτησία τους ε, ταυτόχρονα. Έχετε δύο λεπτά να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όταν μιλάμε για την ε, συνεκτικότητα, τη συνέπεια του Γενικού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων, οι εποπτικές αρχές ε, έχουν το ρόλο να τον εφαρμόζουν. Ταυτόχρονα, ο επόπτης προστασίας δεδομένων ε, έχει και έναν έμεσο ρόλο, ε, ρόλο κλειδί. Είναι και μια μορφή γραμματείας για τον Ευρωπαϊκό Γραφείο Προστασίας Δεδομένων. Επίσης, ως υποψήφιος για αυτή τη θέση, θα ήθελα να ε, υποστηρίξω ένα πρόγραμμα εθνικών ανταλλαγών. Είχα υπηρετήσει και εγώ σε αυτή τη θέση. Η θέση του επόπτη είναι πολύ καλή, γιατί ε, εκεί είναι ο κόμβος για την προστασία των δεδομένων ε, και αυτό σημαίνει πως όταν κανείς βρίσκεται εκεί μπορεί, πρέπει να μιλά μια κοινή γλώσσα μεταξύ των εθνικών αρχών και του Ευρωπαίου Εποπτή Προστασίας Δεδομένων. Εγώ είχα αποσπαστεί ε, στις Βρυξέλλες για έναν τέτοιο ρόλο και αυτό πραγματικά προώθησε την καριέρα μου στην προστασία των δεδομένων. Για μένα ήταν ένας πραγματικός ε, λόγος να εμπλακώ και όταν επέστρεψα στη χώρα μου αυτή η εμπλοκή στο... δραστηριότητε του επόπτη με έκανε πολύ καλύτερο. Ε, φυσικά, Ευρωπαίος Επόπτης παραμένει μέλος του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και έγγραφα και δηλώσεις ε, εκδίδονται βάσει αυτού, όμως για μένα ε, το πιο σημαντικό περιθώριο ε, χειρισμών που υπάρχει είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο και να ανοικοδομηθούν δεσμοί μεταξύ των εθνικών εποπτών και του ρόλου του Ευρωπαίου Επόπτη. Μετά από το το ρόλο έχει η Μπίρκετ Τζίπελ από του Σοσιαλιστές και Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ζάμπο για την εισαγωγή σας. Να επανέλθω στι αγραπτές απαντήσεις σας. Μιλάτε για την έναρξη συζήτηση σχετικά με την αξία ε, των δεδομένων στην οικονομική διαδικασία. Επίσης μιλάτε ε, για το κατά πόσο πρέπει να εξετάσουμε τα στοιχεία της ιδιωτικότητας. Τι σημαίνει αυτό που αναφέρετε, μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα. Επίσης, αναφέρεστε στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιο ρόλο βλέπετε ε, και για το GDPR και για το e στην ανάπτυξη και εποπτεία των αντίστοιχων εφαρμογών ε, τεχνητής νοημοσύνης αν επέλθουν κάποια μέρα. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά για απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ναι, ήταν γενναίο για μένα να αναφέρω τον ε, φόρο ιδιωτικότητας ε, στη γραπτή μου απάντηση. Ε, σε ποιον αρέσουν οι φόροι. Εντάξει, ίσως δεν είναι ο σωστός όρος. Όμως, όταν λέω privacy tax, τι εννοώ. Σκέφτομαι λίγο φωναχτά. Έχω και ακαδημαϊκό υποβαθρό. Νομίζω λοιπόν ότι οι εποπτικές αρχές έχουν την ευθύνη και να εκφράζουν τις ιδέες τους όταν θεωρούν ότι αυτές είναι καλές, να τις ε, αναφέρουν στο κοινό και μετά ε, να συζητιούνται οι ιδέες αυτές. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν αξία και μπορεί αυτή η αξία να εκφραστεί σε ευρώ. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποιούν οι εταιρείε. Ειδικά οι γίγαντες της τεχνολογίας χρησιμοποιούν την ιδιωτικότητά μας ε, και βγάζουν τεράστιο κέρδος. Όπως βλέπω όμως, ε, δεν συνεισφέρουν με σωστό και δίκαιο τρόπο στου εθνικού προπολογισμού. Δεν είμαι ειδικό σε φορολογικά ζητήματα ή ζητήματα προπολογισμού, όμω, όταν σκέφτομαι φωναχτά, θεωρώ ότι ε, με τη χρήση της ιδιωτικότητας μπορούμε και να συνεισφέρουμε στον εθνικό προϋπολογισμό. Λίγο πήρα έπνευση και από τον περιβαλλοντικό νόμο. Τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη και το GDPR και το e-privacy, την ε, εποπτεία του. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι καινούριο σημαίνει ότι σκεφτόμαστε, ε, ότι οι μηχανές σκέφτονται, αλαμβάνουν αποφάσεις και μαθαίνουν. Είναι λίγο τρομακτικό. Η Επιτροπή θα πρέπει μέσα σε, ε, είπε ότι μέσα σε 100 μέρες ε, θα νομοθετήσει γι' αυτό και σε 200 μέρες μας φτάνει. Είναι σημαντικό το θέμα. Ως προς την εποπτεία, το e-privacy και η η εποπτεία των ε, δεδομένων ε, πρέπει να πάνε μαζί. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φέλτε, ένα λεπτό για το Ρινιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σαπο για την εισαγωγή σας. Δεν θα σας ρωτήσω τις απόψεις σας για συγκεκριμένα θέματα, γιατί νομίζω ότι συμμεριζόμαστε τις περισσότερες. Αυτό όμως ε, που έχει να σχέση με τον τρόπο που θα προχωρήσετε ως Ευρωπαίος Επόπτης είναι η ανεξαρτησία και η εφαρμογή κατά δεύτερο λόγο. Ως προς το πρώτο, ξέρουμε ότι ε, ο DPA όπως και ο EDPS συνήθως ε, ε, τίθενται υποπίεση. Στην περίπτωση του Ούγκρου DPA υπήρξε ε, τεράστιος, τεράστια κριτική, για να το πω έτσι λίγο πιο ήπια, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το EDPS λοιπόν πρέπει να είναι και θαραλέος και τελείως ανεξάρτητος δεν έχουμε τους καλύτερους νόμους προστασίας δεδομένων, αλλά η εφαρμογή είναι αυτή που πάσχει περισσότερο. Για το GDPR βλέπω τεράστια πρόστιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Facebook και εδώ πολύ έτσι κυρώσει. κυρώσεις. Πώς θα το αλλάξετε αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Τσαπό δύο λεπτά για την απάντησή σας. Ευχαριστώ κυρία Αντεφέλτ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη. Αν ήμουν στη θέση σας αυτό θα συζητούσα για την ανεξαρτησία και για την Ουγγρική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, DPA. Υπήρξε μια μεγάλη παραβίαση των δεδομένων εκεί και υπήρξε η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Ε, έκλεισε η διαδικασία, τώρα πια δεν συνεχίζεται. Όταν μιλάμε για την ανεξαρτησία, έχω μια έμεση προσέγγιση. Η DPA της ε, Ουγγαρίας, για παράδειγμα, εάν ε, δεν συμμορφώνεται με αυτή την ανεξαρτησία, τότε θα πρέπει η Κομισιόν ως ε, θεματοφύλακας των συνθήκων να παρέμβει και να ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση. Αυτό είναι το νομικό μου επιχείρημα για την πρώτη σας ε, ερώτηση. Τώρα, για την εφαρμογή. Όντως, είναι κομβική σημασία αν έχουμε τους κανόνες και δεν εφαρμόζονται, παραμένουν κενό γράμμα. Η Εθνική, Αρχή, η Εθνική Εποπτική Αρχή μας έδειξε ότι μαθαίνουμε το GDPR κατά κάποιο τρόπο. Όταν ξεκίνησε, κάπως είχαμε απογοητευτεί. Δεν είχαμε ε, δυνατότητες να πάμε διανοσύνοριακά. Ε, χρειάστηκε χρόνος για να μπουν στα μετρό μας υποθέσεις. Όμως σιγά σιγά πολλές αποφάσεις, ακόμα και μεγαλύτερες, ε, θα έλθουν. Ναι, όντως, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ αυστηρές ε, ως προς την επιβολή του νόμου και τη ζηλεύουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγώ λέω ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις. Όμως και μια ξεκάθαρη στρατηγική για την εφαρμογή. Θα προσπαθήσω να προωθήσω αυτό. Τώρα, εκ μέρου των Πρασίνων, ο κύριο Μπράιερ. Είχαμε συναντηθεί πρόσφατα και ένα από τα θέματα που συζητήσαμε είναι ο ρόλος της συγκεκριμένης αρχής. Είχατε πει ότι το EDPS θα πρέπει να δίδει νομικές συστάσεις και να μην κάνει πολιτικές παρεμβάσεις. Έχει όμως ένα συμβουλευτικό ρόλο το EDPS και στην ομοθετική διαδικασία. Μπορείτε να εξηγήσετε λίγο ποιος είναι ο ρόλος που πιστεύετε ότι πρέπει να έχει. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική πώς βλέπω το συμβουλευτικό ρόλο του EDPS. ο σχολιασμός της νομοθετικής διαδικασίας είναι συμβουλευτικός βασικός ρόλος και θα είναι βασικός στόχος των δραστηριοτήτων μου. Είχα πει ιδιωτικά και λέγω και τώρα δημόσια ότι η αρχή αυτή δεν θα πρέπει να, ε, εγγράφεται σε πολιτικό πλαίσιο και να κάνει παρατηρήσεις και σχόλια ε, για θέματα πολιτικής φύσης. Οι γνωμοδοτήσεις και οι απόψεις της συγκεκριμένης αρχής θα πρέπει να είναι αυστηρά νομικής φύσεως. Οι γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να ε, δράζονται στο πρωτογενές και στο δευτερογενές δίκαιο. Ως υποψήφιος ε, βλέπω ότι εσείς ασκείτε πολιτική και το κάνετε καλά. Ε, <clears throat> ευχαριστώ και για τα συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Εγώ κάνω εφαρμοσμένη αν θέλετε πολιτική και ε, γι' αυτό ακριβώς κάνω την διάκριση αυτή που είχα κάνει παλιά ιδιωτικά και τώρα δημόσια. Δεν θα πρέπει ως ε, οργάνωση, ως υπηρεσία να ασχολείται με θέματα πολιτικά. Για την ID, κυρία Τζαρντίνο, ο τομέας των <clears throat> δικαιωμάτων στον τομέα το ψηφιακό. Δώστε ένα δευτερόλεπτο για να μπορέσει να φορέσει τα ακουστικά του. Τα ψηφιακά δικαιώματα είναι κάτι νομικά δεσμευτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις της καινοτομίας μη χάνοντας όμως από τα μάτια της ε, τον κεντρικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων των πολιτών. Εσείς έχετε εμπειρία σε πρακτικό και διοικητικό επίπεδο και μάλιστα ετοιμάζετε και ένα ερευνητικό διδακτορικό, αλλά στον τομέα της προστασίας δεδομένων και των πολιτικών δικαιωμάτων δεν βλέπω να έχετε κάνει κάτι ε, μήπως θα ήταν η στιγμή να βρούμε τη σωστή υπηρεσία ανάμεσα στα δικαιώματα από τα μία και την προστασία των δεδομένων από την άλλη, όπως επίσης <clears throat> και θα ήθελα να μου πείτε αν στα πλαίσια της αυξημένης παρουσίας της τεχνητής νοημοσύνης, αν θα πρέπει η εμπειρία σας να προσφέρει αξία στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πράγματι ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο όλο και περισσότερο και όταν μιλάμε για δικαιώματα αναφερόμαστε και σε ψηφιακά δικαιώματα και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε συνεχώς σε επαφή με τα πανεπιστήμια, με τις ε, ερευνητικέ δραστηριότητες. Αυτό είναι κάτι που αποτελεί προστιθέμενη αξία από το παρελθόν μου Έχουμε ασχοληθεί με πρακτικά θέματα σχετικά με την τεχνολογία και την ιδιωτικότητα. Αν δεν τα συνδυάσουμε αυτά στο θέμα των blockchain σαν παράδειγμα, ε, πώς θα δουλέψει κανείς αν δεν ξέρει τι είναι, ή η τεχνολογία η λεγόμενη hash. Όλα αυτά είναι θέματα τεχνικά και θα πρέπει η αρμόδια αρχή να μην παραπλανηθεί από ελεγκτούς, ελεγκτές συγγνώμη, λέγοντας ότι οι τεχνολογίες χάσουν είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώ είναι πάντα απόλυτα κρυπτογραφημένο. Εμείς θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τον τρόπο λειτουργίας να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και εξελίσσεται και έτσι θα μπορέσουμε να σεβαστούμε ε, τα ψηφιακά δικαιώματα. Σας ευχαριστώ κύριε Τσάμπορ. Ε, ECR Κάνκο. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα είναι σημαντική για τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνικής, τεχνητής νοημοσύνης. Πώς μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε σωστά τις αρχές του EDPR και πώς μπορούμε να ενημερώσουμε σωστά τον πολίτη να ελέγχει τα προσωπικά του δεδομένα στα πλαίσια μιας συνεχούς εξέλιξης, ανάπτυξης ε, της καινοτομίας έτσι ώστε να ξαναγίνουμε ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημαντικό και για τις επιχειρήσεις μας, σημαντικό και την ασφάλειά μας. Όποιος κερδίσει τον πόλεμο του ΆΗ θα κερδίσει και την παγκόσμια οικονομία. Και συνεχίζουμε εμείς να μαθαίνουμε ε, τα πράγματα γύρω από το EDPR. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας σε σχέση με τα μεταδεδομένα, τα metadata. Έχω κάνει μια ανακοίνωση στο παρελθόν. Είναι ένα δύσκολο θέμα γιατί δεν αναφερόμαστε στην ουσία στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Είναι ένα περίπλοκο θέμα αν δείτε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζονται τα μεταδεδομένα, θεωρητικά θα πρέπει να είναι ε, ε, τα στοιχεία του καθενός απόλυτα ε, ορατά καθ' όλη τη διάρκεια της αποθήκεσής τους. Εδώ τίθεται λοιπόν το θέμα της προστασίας τους. Αναφερθήκατε και στην, στην εκμάθηση του GDPR. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσουμε τεχνικές δυνατότητες όλοι, αλλά θα μπορέσουμε να πετύχουμε ε, τον συνδυασμό της υψηλής ε, ταχύτητας των GDPR μέσα από μια μεταβατική περίοδο. Στην πρώτη φάση δεν είχαμε αναμεταδότες. Χρειάστηκα ε, χρόνος για να αποκτήσουμε τους πρώτους αναμεταδότες. Αν σας κατάλαβα καλά, θέσατε ερωτήσεις και σχετικά με την απώλεια ε, των πλεονεκτημάτων τα οποία είχαμε στον τομέα της ε, τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ τίθεται το θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι δεν ελέγχουμε αυτό για το οποίο μιλάμε και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πυκνώσουμε τις συζητήσεις και τότε μόνο ο νομοθέτης θα είναι σε θέση να νομοθετήσει σωστά και τότε μόνο θα υπάρξει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν οι επιχειρήσεις. Για την Γκουε Ντέιλι. Ευχαριστώ. Θα γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα κίνημα προς την διαλειτουργικότητα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων στον τομέα της άμυνας, ασφάλειας, PNR ε, και ε, με πρόσχημα την ασφάλεια. Εσείς πώς ε, αξιολογείτε την κατάσταση σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής και προστασίας δεδομένων υπό το φως των λόγων επιτήρησης που προβάλλονται, που νομίζω ότι προς τα που πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι δεν βλέπετε το ρόλο σας ως πολιτικό ρόλο, αλλά η επιτήρηση είναι πολιτικό θέμα και νομικό θέματα και το δικαστήριο έχει ήδη κάποια νομικά μέσα. Πώς βλέπετε εσείς το ρόλο σας εδώ, γιατί δεν νομίζω να είναι απλά νομικός και ορισμένες πτυχές έχουν ήδη εντοπιστεί ότι δεν συμβαδίζουν με το, τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Ζάμπο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Πράγματι, κάποιες φορές είναι παραπλευνητικό να σκέφτεται κανείς ε, τα νομικά θέματα ότι δεν έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Θυμάμαι όταν ήμουν νεότερος και δικηγόρος, νέος δικηγόρος είχα κάνει μια τεράστια ε, έρευνα για το CCTV, για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Μετά από χρόνια καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα νομικά, ξεκάθαρα νομικά συμπεράσματα που ε, αφορούσαν την έννοια της νομοθεσίας είναι ένας χαρακτηριστικός τομέας επιτήρησης, ασφάλειας και θεμάτων ιδιωτικότητας, ιδιωτικής ζωής. Αυτά για το γενικό πλαίσιο. Τώρα, στη διαλειτουργικότητα, βεβαίως η αρχή προστασίας δεδομένων το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων μας θυμίζει για τις αρχές που διέπουν αυτό το πλαίσιο. Ε, επίσης, το γεγονό ότι οι συνομοθέτε έχουν ε, περάσει ένα νόμο για βάσεις δεδομένων όπως θέματα διαφάνειας που δεν είναι εναντίον της ασφάλειας. Επίσης, να θυμηθούμε ότι Εάν γίνει πραγματικότητα η λειτουργικότητα, τότε ο εποπτικός ρόλος μας θα είναι πιο περίπλοκος. Θα είναι πιο δύσκολο να εποπτεύεις ε, μια τόσο περίπλοκη ανταλλαγή δεδομένων. Για μένα το κλειδί είναι εδώ. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή. Και αυτή είναι μια συνεχής προσπάθεια των αρχών προστασίας δεδομένων. Για τους ενάει η κυρία Φόξ. Κύριε ο κανονισμός GDPR είναι για την προστασία των ε, ε, δεδομένων, ε, αλλά είχε αρνητική επίδραση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε φιλοανθρωπικούς οργανισμούς και στην κοινωνία των πολιτών γενικά. Ε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οι μεγάλες πολυεθνικές με στρατώνες που τα βάζουν με μικρού οργανισμού που προσπαθούν να έχουν επαφή με τα δίκτυά τους και να κτίσουν στήριξη ανάμεσά τους και αντιμετωπίζουν ε, τις ίδιες κυρώσεις, ε, δρακόντιες κυρώσει, Έχει δημιουργηθεί έχουν δημιουργηθεί θέσεις ε, εργασίας για, για τον έλεγχο αυτού του κανονισμού. Πώς μπορείτε να μου διασφαλίσετε ότι η προστασία της ιδιωτικότητα δεν οδηγεί σε υπέρμετρη ρύθμιση και κανονισμό και δεν στραγγαλίζει την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, αρνείται την ελευθερία σε μικρούς οργανισμούς μικρομεσαίους και στην κοινωνία των πολιτών να λειτουργήσει. Κύριε Ζάμπο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Όταν ήταν ακόμα σε στάδιο προσχέδιο GDPR, ένα από τα κύρια μηνύματα ήταν να αποφύγουμε το επιπρόσθετο διοικητικό άχθος. Αυτό ήταν κάτι το οποίο προσπάθησαν πάρα πολλοί νομοθέτες να πετύχουν και αναφέρεται πράγματι ε, στο γενικό πλαίσιο του κανονισμού GDPR. Θέλω να πω ότι η αξιολόγηση συνεχίζεται του κανονισμού αυτού και είμαι βέβαιος ότι αυτή η πτυχή του επιπρόσθετου διοικητικού άχθους θα είναι μία από τις πτυχές που θα ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή. Τώρα, όταν μιλάμε για μικρούς οργανισμούς, αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ε, μικροί, οργανισμοί στο να ε, υλοποιήσουν τον κανονισμό GDPR. Πρέπει να πω ότι η, αρχή, η Ουγγρική Αρχή Προστασίας των Δεδομένων και άλλες αρχές έχουν κάποια προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν μια γραμμή, τηλεφωνική γραμμή δική που μπορούν να καλούν και μπορούμε να απαντούμε ερωτήσεις ε, και απαντούμε και στις ανησυχίες τους και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή του GDPR και θα δημοσιεύσουμε ε, κάποια αποτελέσματα σε ένα έγγραφο. Θα παραμείνει στόχος η μείωση του διοικητικού άχθου, άχθους για, τις, ε, για τον νομοθέτη και τις αρχές. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Επανερχόμαστε στον κύριο Λένας από πλευρά ΣΕΛ και ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πράσινοι ρώτησαν ακριβώ την ερώτηση που ήθελα εγώ να υποβάλω. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα. Βέβαια, μπορεί να περνάμε διαφορετικέ απαντήσει, αλλά απαντήσατε σαφώ ε, για το θέμα του GDPR. Ίσως θέλετε να αναπτύξετε για το πώς θα διασφαλίσετε ότι το EDPS υπό την εποπτεία σας θα δει στην πράξη αυτή την εφαρμογή. Τώρα για τη διαλειτουργικότητα νομίζω έχουμε βρει τη χρυσή τομή. Ε, είπατε ότι θα είναι πιο δύσκολο για σας να αναλάβετε τον εποπτικό σας ρόλο στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας. Θα μπορούσατε να μας πείτε ακριβώς ποια θα είναι η προσέγγιση σας τα επόμενα χρόνια όταν θα είμαστε στην εφαρμοστική φάση ε, έτσι ώστε το EDPS να είναι έτοιμο να αναλάβει τον εποπτικό ρόλο ακόμη ε, ε, και με την διαλειτουργικότητα. Κύριε Ζάπο, δύο λεπτά για την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ε, νόμιζα θα με υποβάλλετε δύο φορές την ίδια ερώτηση. Χαριτολογώντας. Τώρα για τη διαχωρισμό των δύο ρόλων. Αν μιλάμε για την επιβολή ή την παροχή συμβολών ή το νομικό και τον πολιτικό λόγο, πιστεύω, ρόλο, πιστεύω είναι σαφές. Οι αρχές εποπτείας ε, δεδομένων έχουν να κάνουν με το νόμο για την προστασία των δεδομένων. Και πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος. Πρέπει να ξέρουμε Ποιο έχει το ρόλο της λήψη αποφάσεων στην πολιτική, στην νομοθεσία και ποιο έχει το συμβολευτικό ρόλο ως αρχές εποπτείας ε, δεδομένων. Για μένα, ως επικεφαλής ενός ε, τέτοιου γραφείου, δεν είναι δύσκολο να διαχωρίσω αυτούς τους δύο ρόλους. Ε, ρωτήσατε και για την εποπτεία και την διαλειτουργικότητα. Εάν το σύστημα ξεκινήσει να λειτουργεί και θα γίνεται ανταλλαγή ε, προσωπικών δεδομένων ως καθημερινή ρουτίνα. Βέβαια, η εποπτεία δυσχεραίνεται. Είναι πιο περίπλοκος ο ρόλος μας εδώ, γιατί πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές ε, εποπτείας και το NDPS. Έχουμε ε, την εθνική πτυχή και την κεντρική πτυχή όλων αυτών των ανταλλαγών δεδομένων. Αυτό που κάνουμε και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που τερέχει στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων είναι να βελτιώσουμε ε, τους τρόπους μετάδοσης και βλέπω χώρο ε, όπου μπορούμε να κάνουμε πιο ε, αυστηρά αυτά τα όρια και να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο εποπτείας. Ευχαριστώ κύριε Ζάμπο. Άλλο ένα λεπτό. Η σειρά σας κύριε Μωράης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω και η δική μου ερώτηση καλύφθηκε, αλλά ε, θα την ε, κάνω με άλλο τρόπο. Ο συμβουλευτικός ρόλος σας. Αυτό που μαθαίνουμε από το EDPS είναι ότι έχετε πολλά ε, στοιχεία στην εντολή σας που έχουν να κάνουν με την παροχή συμβουλών στην Κομισιόν, όμως αυτή μπορεί να σας αγνοήσει αν εσείς κάνετε μια πρόταση. Αυτός είναι ένας πολιτικός ρόλος. Τι θα κάνετε αν αποφασίσει η Επιτροπή να σας αγνοήσει. Και μετά αναφέρετε το Cambridge Analytica. Όλοι οι υποψηφοί θα αναφέρουν αυτή την υπόθεση. Υπάρχει όμως ένας πολλαπλασιασμός ε, μεθόδων, ε, εφαρμογών που χρησιμοποίησαν ε, και υπήρξε νοθεία των εκλογών με αυτόν τον τρόπο, ε, στην μια μορφή νοθείας των εκλογών με αυτόν τον τρόπο. Εσείς πώς θα θέσετε προτεραιότητες και πώς θα αντιμετωπίσετε αντίστοιχα ζητήματα. Παρακαλώ, η απάντησή σας κύριε Ζάπο. Ευχαριστώ. Δύο περίπλοκα ζητήματα θέσατε βασικά. για την επικοινωνία με την Επιτροπή. Ο Ευρωπαίος Εποπτής Προστασίας Δεδομένων κάνει κάποια σχόλια και αυτά γνωρούνται. Αυτή είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο Επόπτης έχει λάβει θέση και είναι πια ε, κομμάτι της κουλτούρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Εγώ θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια να επαναλάβω τα όσα λέω να ακουστεί η φωνή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό λοιπόν ο επόπτης να δρά ως σύμβουλος και ο CDPS μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη θέση για ένα θέμα, αλλά είναι σύμβουλος. Με κάθε σεβασμό λοιπόν και σε στενή επικοινωνία, αλλά ο σύμβουλος πρέπει να αποδεχτεί αν αγνοηθεί. Κατά τη διάρκεια βέβαια της νομοθετικής διαδικασίας ε, πρέπει να είναι διαθέσιμος για όλα τα θεσμικά όργανα και του συνομοθέτες με επίσημο και άτυπο τρόπο. Ω σύμβουλος όμως κάποιες φορές αντιμετωπίζει αυτό το θέμα να σε αγνοούν. Τώρα, για το Cambridge Analytica. Αναφέραμε σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες τεχνολογίες, γιατί αυτό που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του σκανδάλου, που δεν ξέραμε τι συμβαίνει, ήταν αυτή η παγίδα των αόρατων δεδομένων, όχι μόνο αποφάσεις, ε, ε, διαδικασίες επεξεργασίας που είναι αόρατες. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο μας να παρακολουθούμε τις νέες ε, τεχνολογίες, να υπάρχει συνεργασία και να συλλέγουμε στοιχεία για τα συνεχώς αναδυόμενα θέματα. Η συνεργασία νομίζω είναι το κλειδί. Ευχαριστώ. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους ευρωβουλευτές που έκαναν ερώτηση. Ευχαριστούμε ειδικά τον κύριο Ζάμπο, όχι μόνο για τις απαντήσεις σας, αλλά Επιμένω και για το γεγονός ότι τα καταφέρατε να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι αυτό το στάδιο, στην Επιτροπή μας, που θα αποφασίσει αύριο. Όπως και να έχει, έχετε δύο λεπτά για την τελική σας δήλωση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν πολύ καλή η συζήτηση μαζί σας. Πραγματικά χάρηκα που συζητήσαμε για την προστασία των δεδομένων και τα ζητήματα της ιδιωτικότητας. Απήλωσα την συζήτηση, ακόμα και αν ερωτήσεις, κάποιες ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν στο πλήρε εύρο τους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Βλέπω μεγάλες συνέργειες στη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι θέσει του θα παραμείνουν ω έμπνευση για το μέλλον. Τώρα πρέπει να σας χαιρετήσω. Ε, ως ε, εκπροσώπους ε, των πολιτών μας για λιγάκι και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα στο προσεχές μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζάμπο. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τώρα δεν χρειαζόμαστε άλλη εισαγωγή ως προς τη μέθοδο, γιατί τη μάθαμε. Θα είναι και πάλι πέντε λεπτά για τον κύριο Βερόφσκι, τον οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί είχε αυτή τη θέση τα τελευταία πέντε χρόνια ως ε, βοηθός ε, στον Ευρωπαϊκό Προστασία Δεδομένων. Και πάλι θα έχουμε δέκα ερωτήσεις στον δεύτερο αυτό υποψήφιο για τη θέση του Ευρωπαίου Εποπτή Προστασίας Δεδομένων, ή e DPS. Ένα λεπτό η κάθε ερώτηση, δύο λεπτά η κάθε απάντηση και μετά η τελική δήλωση δύο λεπτά. Έχετε το λόγο Καλώς ήρθατε. Αφήστε με, όμω πριν από όλα αυτά, να σας ε, συγχαρώ όχι μόνο που θέσατε υποψηφιότητα, αλλά και που καταφέρατε να επιλεγείτε από την Επιτροπή ε, Επιλογών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και να φτάσατε στο στάδιο να ψηφίσει αύριο η Επιτροπή μας για την υποψηφιότητά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα που είμαι ανάμεσά σας και σας παρουσιάζω το όραμά μου και τις προσδοκίες μου για τα επόμενα χρόνια στα πλαίσια της προστασίας δεδομένων, της προστασίας της ιδιωτικότητας και του ε, επιβλέποντος την υπηρεσία αυτή. Θα προσφέρω ότι περνάει από τα χέρια μου θα προσφέρω τις αξίες, την εμπειρία, τις γνώσεις. Πριν πέντε χρόνια ήμουν πάλι παρόν εδώ, υποψήφιος για τη θέση του βοηθού και προερχόμαι από μια χώρα η οποία ήταν ολοκληρωτική πριν από το 1989 και οι αξίες αυτές μας είχαν λείψει για πάρα πολύ καιρό. Έχω όμως και την εμπειρία νομίζω που χρειάζεται και από τον ιδιωτικό τομέα στον οποίο δούλεψα για 7 χρόνια και δεν είμαι απλά ένας δικηγόρος που προετοίμαζα συμβάσεις, αλλά έκανα την επιμελητία, έκανα το λεγόμενο data mining, την εξόριξη των δεδομένων και νομίζω ότι απέκτησα την κατάλληλη εμπειρία. Εργάστηκα επίσης και σε δημόσιες υπηρεσίες και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων σε διεθνές επίπεδο. Έχω λοιπόν συνολικά 25 χρόνια εμπειρία σε πανεπιστημιακό επίπεδο και γι' αυτό ακριβώς τεχνολογικά είμαι σε θέση να κατανοώ τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας και γνωρίζω πώς λειτουργεί φυσικά η υπηρεσία, πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά όργανα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και πού τα πράγματα είναι θετικά ή αρνητικά. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα επόμενα λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας. Πέντε είχατε συνολικά. Καλά, λίγα επιπλέον λόγια λοιπόν. Η εμπειρία από τη μία είναι θετική, από την άλλη υπάρχει αν θέλετε και μία αντιμετώπιση των προβλημάτων της προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικότητας και σε επίπεδο ηλικιακό. Είμαι με 40 χρόνια νεότερος από τον προηγούμενο, αλλά ξεκίνησα εγώ να χρησιμοποιώ υπολογιστές όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο και έχω και δύο κόρες οι οποίες είναι θα έλεγα γηγενείς του ψηφιακού κόσμου. Συνεπώς λοιπόν πιστεύω ότι ο κόσμος αυτός μπορεί να διατηρήσει τις αξίες μας και να χρησιμοποιήσει τις καινοτομίες με σωστό τρόπο έτσι ώστε ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ευχαριστώ τον κύριο Βεβερόσκη και θα ακολουθήσουν δέκα εν σειρά του ενός λεπτού η καθεμία και δύο λεπτά για την απάντηση. Όλα. Ε, σας ευχαριστώ στα πλαίσια της εμπειρίας σας ως ε, βοηθού διευθυντή του EDPS. Πώς βλέπετε εσείς η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώνει τις αποδόσεις της στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων σε συνεργασία με μη κοινοτικού παίκτες, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων και την καινοτομία γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να προστατευτούν τα δεδομένα και των Ευρωπαίων και σε συνεργασία με μη ευρωπαϊκούς παίκτες. και ε, υπάρχει δυνατότητα χρήσης ε, των πνευματικών δικαιωμάτων θα έλεγα και της νομοθεσίας τους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κοιτάξτε σε δύο λεπτά είναι δύσκολο να απαντήσω γιατί συνδυάζονται πάρα πολλά πράγματα στην ερώτησή σας. Θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα υπέρ Τη συζήτηση για την ιδιοκτησία των δεδομένων και την ιδιοκτησία κυρίως των στοιχείων ενημέρωσης. Εγώ σαν δικηγόρος έχω την εμπειρία που μου παρέχει το αστικό δίκαιο ε, που έχει κανείς την δυνατότητα να πωλήσει κάτι, να μοιραστεί κάτι, να εγκαταλείψει κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να δουλέψει με τα δεδομένα. Αν θέλει κανείς να ελέγξει τα δεδομένα, σημαίνει ότι οι μοναδικοί που μπορεί να μεταχειριστούν, να χειριστούν τα δεδομένα είναι αυτοί οι οποίοι τα καταθέτουν. Συνεπώς και όσο πιο περίπλοκο γίνεται το σύστημα, όλο και πιο δαλειτουργικά καθίστανται τα συστήματα, τόσο πιο περίπλοκοι και σύνθετοι είναι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται. Αν σκεφτούμε τώρα λίγο το θέμα της αντιμετώπισης των εμπλεκομένων στην αγορά και όσων ασχολούνται με θέματα ιδιωτικότητας εδώ θα ήθελα να τους διαιρέσω σε τέσσερις ομάδες. Κράτος, διεθνείς οργανισμοί, διεθνή φόρα, διαφορετική αντιμετώπιση του επιχειρηματικού κόσμου και διαφορετική αντιμετώπιση της κοινωνίας των πολιτών και τα τέσσερα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, σχετικά με το κράτος και τα διεθνή φόρα θα ήθελα να υπογραμμίσω σε επίπεδο ε, ε, μετά από τις τελευταίες ρυθμίσεις στη συνέργεια ανάμεσα στις υπηρεσίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους υπόλοιπους εταίρους στον χώρο του κράτους. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς το κάνουμε αυτό. Έχουμε δημιουργήσει το λεγόμενο Hack Forum. Εμείς συζητάμε τα θέματα των συμφωνιών με παρόχους υπηρεσιών εκτός ε, δημοσίου και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Δεδερός και προσπαθήστε παρακαλώ να μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, η εκπρόσωπος ε, του, ε, των σοσιαλιστών κυρία Ζήπελ. Σας ευχαριστώ κύριε Βιμπερόφσκι, σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας σχετικά με την ιδιοκτησία των δεδομένων και εκεί έχουμε κάποιες αντιρρήσεις. Στη δήλωσή σας αναφερθήκατε και στην πρόκληση που έχουμε για τη διατήρηση των αξιών μας. Πώς εσείς βλέπετε τον ρόλο του GDPR και της προστασίας της ιδιωτικότητας στον τομέα της ανάπτυξης του ελέγχου ε, των ε, εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπονται νέα μέτρα, είναι απαραίτητα, πρέπει να γίνουν συζητήσεις γύρω από αυτά σχετικά με την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Και μια δεύτερη ερώτηση ε, ο κανονισμός ε, e-privacy δεν πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα. Εσείς βλέπετε ότι θα υπάρξει δυνατότητα να πιέσουμε για μια πιο έντονη και σωστή εφαρμογή ε, των ισχυουσών διατάξεων μεταξύ των οποίων και τα λεγόμενα cookie rules, όπως επίσης και τις ε, ανιχνεύσεις προσώπων μέσω του διαδικτύου. Βέβαια, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας. Είναι πρόκληση για τις αρχές προστασία των δεδομένων, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα τι εννοούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας όρος marketing, μια έννοια marketing που μπορεί να συνίσταται ε, σε, σε ρομποτική, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και για την αναγνώριση προσώπου, η fake news, που είναι διαφορετικά θέματα, που είναι και σημαντικά, πρέπει να συζητηθούν μεν, αλλά όχι κατά ανάγκη στο πεδίο εφαρμογή ε, της τεχνητή νοημοσύνης. Αυτό που πιστεύω ε, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε τι έχουμε στη διάθεσή μας, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο κανονισμός GDPR είναι μία από τις νομοθετικές παράξεις που μπορεί να καλύψει ή να έχει πολλές προσδοκίες ε, προς τον κανονισμό της τεχνητής νοημοσύνης Ταυτόχρονα πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα μέρη που δεν ρυθμίζονται σωστά και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των αλγορίθμων που ε, δεν καλύπτονται κατά ανάγκη από τον κανονισμό GDPR. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ήδη έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες σε πολλές χώρες σχετικά με τα συστήματα κανόνων που δεν είναι τεχνητής νοημασίνης αλλά που θέτουν τα ίδια προβλήματα που είχαμε και στην τεχνητή νοημασύνη. Και δεν έχουμε απλά την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση του πώς έχουν γίνει αυτά. Σχετικά τώρα με το e-privacy. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει ε, με αυτό την ε, συζήτηση γιατί έχει δοθεί γνωμοδότηση για τι τρέχουσε σχέσεις ανάμεσα ε, στο e-privacy και το GDPR, αλλά ταυτόχρονα το πρόβλημα που αγγίξατε των cookies, ιδιαίτερα των cookie walls, που είναι μια πρόκληση για την εναρμονισμένη προσέγγιση στην Ευρώπη, ειδικά γιατί οι αρχές προστασίας δεδομένων δεν είναι πάντα υπεύθυνε για αυτό το μέρος. Ε, ευχαριστώ. Renew, η κυρία Σοφία Ιντεβέλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Βιβερόφσκι. Χαιρετίζω την προσωπική σας δέσμευση, από την βαθιά σας πεποίθηση και νομίζω συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Ωστόσο, αυτός ο διορισμός δεν ε, αφορά μόνο τις απόψεις σας. Έχει να κάνει και με το πώς εσείς θα κάνετε θα δώσετε περισσότερη δύναμη ε, στην αρχή εποπτείας προστασίας των δεδομένων, διότι ε, μερικές φορές φαίνεται να είναι ένας τυπικός ρόλος ε, και τον οποίο αγνοεί η Ευρώπη εις βάρος της ιδιωτικότητας και η Κομισιόν ήδη έχει χάσει πολλές υποθέσεις στο δικαστήριο, PNR, η privacy ασφαλών λιμένων τι θα κάνετε εσείς για να δώσετε περισσότερη δύναμη στο EDPS και θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι η οδηγία, η λεγόμενη Police ε, Directive θα αντικατασταθεί από κανονισμό. Δύο λεπτά κύριε Βιβρόσκη. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξουμε την ισχύ του EDPS πιέσει μέσα από την επιβολή και την ε, ε, εφαρμογή των κανόνων που έχουμε στα χέρια μας, να δείξουμε ότι υπάρχει ε, λόγος ε, να δοθεί δυνατότητα στις αρχές προστασίας δεδομένων να ασχολούνται με τα θέματα ε, που ανατίθενται από το Κοινοβούλιο, ε, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα δώσω έμφαση στην πρακτική δουλειά που γίνονται, γίνεται από τους θεσμούς συμπεριλαμβανομένου EDPS. Θα ήθελα να τονίσω επίσης κάτι άλλο σημαντικό. Είναι ότι θα πρέπει να βγούμε εμείς ως EDPS και θα βγούμε, να βγούμε από το νομικό πεδίο συμβουλών, να δίνουμε τεχνικές συμβουλές ε, στους θεσμούς. Είναι κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό αποφασίσαμε τον τελευταίο μήνα να έχουμε τον πρώτο <clears throat> επιστήμονα ε, που ασχολείται με τα δεδομένα στον οργανισμό μας και ο τελευταίος διαγωνισμός που είχαμε ε, έχουμε δώσει περισσότερη έμφαση στη διαφορετικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, διότι η διαφορετικότητα στο, στο γραφείο θα είναι ε, σημαντικό για να δώσουμε ακριβώς αυτό που περιμένετε από εμά, όχι μόνο την νομική ανάλυση, αλλά και την πρακτική συμβουλή. Αυτό θα είναι το σημαντικότερο ίσως για να ε, παραμείνει ο, ρόλος μας, ο συμβουλευτικός μας ρόλος προς τα θεσμικά όργανα. Ποιο ήταν το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Θα συμφωνούσατε ότι η λεγόμενη πολύ ε, ε, αστυνομική οδηγία α, την πρώτη φορά, στην πρώτη συνάντηση της ΛΥΠΕ το 2012, είχα την ευκαιρία να μιλήσω ακριβώς για αυτή την οδηγία που λέει ότι είναι μια συνεκουανών προπόθεση να δοθούν στις αστυνομικές αρχές το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία για τα μεγάλα δεδομένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κανονισμός αυτή η οδηγία, αλλά θέλω να δω μια οδηγία που τουλάχιστον να έχει την όψη ενός κανονισμού. Ευχαριστώ. Η πράσινη για ένα λεπτό. Κύριος Μπράιερ. Ευχαριστώ. Κύριε Βεροσκή, ευχαριστούμε πολύ για την ε, υποψηφιότητά σας ε, και βέβαια ε, δεν είναι εκπληξή που έρχομαι εδώ με μια ερώτηση για τα δεδομένα ε, τοποθεσίας και την μη διάκριση και την κράτηση όλων των δεδομένων κυκλοφορίας και τοποθεσίας. Φαίνεται πως η τήρηση τέτοιων δεδομένων δεν είναι ανάλογη προς την ανάγκη πάταξης της τρομοκρατίας. Ε, το προσωπικό στην υπηρεσία σας είπε ότι ίσως ο υπόπτης μπορεί να έχει μια ε, μικρότερη αλλά αποτελεσματική διατήρηση αυτών των ε, δεδομένων σε συμφωνία με τη χάρτα. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση για αυτό το θέμα, ε, η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε κατά τέτοιων ας πούμε δράσεων που εφαρμόζονται σε όλο τον πληθυσμό έτσι στα τυφλά. Η πολιτικές σας. Πώς θα μας υποστηρίξουν σε αυτό το επίπεδο. Κοιτάξτε, θέλουμε ίση μεταχείριση σε όλους τους ε, υποψηφίους. Παρακαλώ, ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση. Να μείνετε πιστοί σε αυτό. Κοιτάξτε, στον ιδανικό κόσμο δεν θα ήθελα να βλέπω την κράτηση προσωπικών δεδομένων δεν θα ήθελα να υπάρχει καμία δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα επίσης που κρατούνται, διατηρούνται για τεχνικούς λόγους. Την ίδια στιγμή όμως, όντως, όντας σύμβουλο σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπηρεσίες αλλά και στους νομοθέτες πρέπει να λάβω υπόψη και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά και την τρέχουσα κατάσταση. Και αναρωτιέμαι, η κατάσταση που έχουμε τώρα που δεν έχουμε οδηγία για την ε, διατήρηση και κράτηση δεδομένων και δεν έχουμε απαγόρευση, γιατί δεν έχουμε απαγόρευση, είναι σωστή αυτή η κατάσταση. έχω, δεν έχουμε λοιπόν αυτή την απαγόρευση και αν έχουμε ένα δικαστήριο που λέει ότι δεν υπάρχει γενικά σύγκρουση μεταξύ του εις ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και της κράτησης δεδομένων, αλλά θέτει ένα ανώτατο όριο πολύ αυστηρό, εγώ το όριο θα κοίταζα. Αυτό το κατόφλι. Δεν θέλω να, γενικά να έχουμε τήρηση τέτοιων δεδομένων, όμως με τις ε, καταστάσεις και τις λύσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε διαφορετικοί από χώρε που δεν έχουν καθόλου τήρηση τέτοιων δεδομένων και από αυτές που έχουν ως τακτική διαδικασία να ε, ψάχνουν στις τηλεπικοινωνίες για να βρουν τέτοια στοιχεία και να τα διατηρήσουν. Άρα, θα ήθελα ε, όταν τα κράτη-μέλη ασκούν πίεση να θυμούνται ότι υπάρχει αυτό το ανατοτόριο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πότε χρησιμοποιείς αυτά τα δεδομένα. Δεν μου άρεσε μια δήλωση ενός ε, επιτρόπου ε, πριν από μερικά χρόνια που είπε ότι η κράτηση δεδομένων ήρθε για να μείνει. Ε, παραδέχομαι όμως ότι από τεχνική και εμπορική άποψη κάπου εκεί βρίσκονται αυτά τα δεδομένα. Άρα για μένα ποιος θα έχει πρόσβαση, πότε και για ποιο λόγο, ποιο σκοπό. Αυτό είναι που μετράει. Ευχαριστούμε κύριε Βερντρόφσκι. Και τώρα για το ID. Βιρτ Ένα λεπτό, όχι καμία ερώτηση. Ωραία, τότε πάμε στην κυρία Κανκό για το ECR. Α, ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ένα γρήγορο στοιχείο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Γιατί στη γραπτή σας απάντηση βλέπω κάτι με το οποίο μπορώ να σχετιστώ. Ε, πώς αισθάνεται κανείς ε, για, μια, για έναν τομέα τον οποίο γνωρίζει καλά. Θυμάμαι την παιδική μου ηλικία. Χαίρομαι πολύ ότι που ο δικτάτορα που είχαμε δεν είχε ίντερνετ, γιατί θα μπορούσε να κάνει περισσότερα στον πληθυσμό μα από ό,τι έκανε. Έτσι λοιπόν σας ζητώ να μου απαντήσετε μια ερώτηση σχετικά με την ζωή του GDPR. Πόσο ε, θα διαρκέσει. Φαίνεται ότι επικεντρώνεται πάρα πολύ ε, σε διατακτικούς κανόνες ε, ε, και ξέρετε ότι η τελευταία νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων κράτησε 20 χρόνια. Επειδή είναι κανονισμό στο GDPR, πόσο νομίζετε ότι θα κρατήσει, θα διαρκέσει. Και ποια είναι τα επόμενα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη φάση. Έχετε το λόγο κύριε Βίβεροφσκι. Αν καταλάβα καλά, η ερώτηση είναι το τι θα πρέπει να γίνει ε, στο μέλλον. Ναι, να σκεφτούμε λίγο πιο πολύ μπροστά, γιατί το GDPR, ε, κοιτάξτε, είναι γιαούρτι που έχει λήξει εδώ και μια εβδομάδα. Κοιτάξτε, για μένα το GDPR δεν είναι η μόνη νομική πράξη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όταν μιλάμε για την Ευρώπη ως ηγέτη στον τομέα της ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων, θα πρέπει να μιλάμε για ολόκληρο το κοινοτικό και εκτιμένο. Δεν είναι θέμα λοιπόν μόνο του GDPR και του e-privacy, είναι ολόκληρο το νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει κάποιο συγκρίσιμο κριτήριο στην παγκόσμια συζήτηση, ένα benchmark. Και αυτό δεν θα μας οδηγήσει σε ε, συνθήκη για την προστασία των δεδομένων στο εγγύ μέλλον. Αλλά θα μας επιτρέψει να μοιραστούμε αξίες με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές χώρες. Ευχαριστούμε. Και τώρα περνάμε στην ΚΟΕ. Ο κύριος Μπαρένα. Σωστά. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Μπαρένα. Uh, uh, Ευχαριστώ. Το άρθρο 61 και 62 του κανονισμού 2018-25 ε, έχει την υποχρέωση συνεργασίας ε, με τις εθνικές αρχές. Είναι μέσα στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία συστημάτων πληροφορι... πληροφορικής ε, μεγάλης κλίμακας ε, και του Eurorack, το Σέγγεν, το σύστημα για τα τελωνία. Μπορούμε να μιλάμε για ώρα, ε, για τα εκατοντάδες εκατομμύρια μάλλον προσωπικών δεδομένων που φυλάσσονται. Ποια είναι λοιπόν η πρόκληση που αντιμετωπίζει ένα συντονισμό τέτοιων ε, δεδομένων, πώς θα διασφαλίσετε την αποτελεσματική εποπτεία αυτών των συστημάτων πληροφορικής, κύριε Φιβρός, και έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Από όσο ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε μυριάδες λύσεις όσον αφορά στην εποπτεία των διοκτικών αρχών αλλά και των διαφόρων βάσεων δεδομένων που υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιπλέον. Η εικόνα αυτών των δεκάδων ε, βάσεων δεδομένων και πόρων ε, που μοιράζονται και ανταλλάσσουν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες. Όλα αυτά μας δείχνουν πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα. Πάντοτε καλούμε για να του όσον αφορά τα συστήματα εποπτείες. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι λύσεις αυτή τη στιγμή στον κανονισμό 17-25 στο κεφάλαιο 9 δεν αρκούν κάποιες φορές ε, έχουμε κάποια πράγματα στην Ευρώπη ε, που είναι πολύ καλύτερα από αυτό. Επίσης υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ των πραγμάτων που γίνονται από τα θεσμικά όργανα όπως ε, η Όλαφ και από τις βάσεις δεδομένων που έχει η Γιουλίζα και από τη συνεργασία που έχει η Eurojust. Κατανοούμε λοιπόν αυτές τις διαφορές και γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή λύση. Ταυτόχρονα να τονίσω ότι όταν μίλησα για επιβολή στον τομέα της προστασίας δεδομένων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τέτοια ε, τέτοιες υπηρεσίες εννοούσα αυτές που ασχολούνται με τις διοκτικές αρχές και τα δεδομένα τους αλλά και τα αστυνομικά δεδομένα. Την περασμένες εβδομάδες είχαμε ένα θέμα με τις πρώτες απαγορευτικές ε, αποφάσεις για αυτό το θέμα. Ας πούμε, απαγόρευση της δραστηριότητας ε, παρακολούθησης των κοινωνικών υπηρεσιών από μία από τις υπηρεσίες που δεν είχε αρκετό νομικό υπόβαθρο για αυτή τη δραστηριότητα. Ε, αυτή δεν ήταν εύκολη απόφαση γιατί κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες, αλλά δυστυχώς χωρίς τη συμφωνία του νομοθέτη δεν πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κύριε Βερόσκη, στα δύο λεπτά να μείνετε παρακαλώ. Και τώρα η ε, κυρία Φόξ ε, για τους ε, μία γραμμένους. Κύριε και μία από τις μεγάλες απειλές για τις ε, πολιτικές ελευθερίες σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα να κρύψουμε, τίποτα να φοβηθούμε. Και τελικά ο φόβος ε, και η επιδίωξη του φόβου είτε μέσω της εθνικής ασφάλειας είτε της κυβερνοασφάλειας που ασκούν κράτη-μέλη, κυβερνήσεις και ευρωπαϊκά ε, σώματα. Αυτά είναι που οδηγούν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και μαζική παρακολούθηση. Ε, οι εταιρείε ε, τεχνολογίας κρυπτογραφούν μηνύματα και υπάρχουν αυτά τα μυστικά μηνύματα κατά του κράτους. Αυτό πραγματικά για μένα είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές. Αναρωτιέμαι λοιπόν ο EDPS ε, τι ακριβώς ε, θα κάνει ε, όταν η εθνική αυτή κατάσκοπη κατασκοπεύουν τους πολίτες τους. Δεν είναι καλό η κυβέρνησή σου να σε κατασκοπεύει. Η απάντησή σας κύριε Μιβερόφσκη. Υπάρχουν δύο μορφές απαντήσεων και δύο ομάδες απαντήσεων. Αν, εξαρτάται αν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια ή για την ασφάλεια Γιατί και τα δύο βάλατε στην ίδια ερώτηση. Ενώ υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ τους, μόνο και μόνο από τυπική άποψη. Εγώ θα ήθελα να βλέπω ένα διακριτό όριο μεταξύ των ε, πραγμάτων που αφορούν στην εθνική ασφάλεια και τα οποία θα πρέπει διαφορετικά να αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και η νομοθεσία και ε, μεταξύ αυτών λοιπόν και της κυβερνοασφάλεια. Θα ήθελα μάλλον να προτείνω λοιπόν ότι αφού συμφωνούμε κάθε χρόνο ε, ότι υπάρχουν νέες μορφές ε, παρακολούθησης που κατά κάποιο τρόπο είναι αποδεκτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το κάνουμε λίγο πιο καινοτόμα και να αφαιρούμε ένα παλιό στοιχείο για κάθε καινούριο που προτείνουμε. Αν κάτι δεν είναι αποτελεσματικό και θέλουμε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο, ας το αντικαταστήσουμε, μην το προσθέσουμε το καινούριο, γιατί όπως περνάει ο καιρός, τελικά ο EDPS ε, φτάνει σε μια κατάσταση που έρχεται στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν και λέει Τώρα μιλάμε για αυτό το βήμα και σε πέντε χρόνια θα επανέλθουμε να μιλήσουμε για ένα άλλο βήμα. Αν τώρα μιλάμε για τη διαλειτουργικότητα, ποια θα είναι η συζήτηση σε πέντε χρόνια. Θα πάμε πίσω. Δεν είναι αστείο αυτό, δεν είναι ανέκδοτο. Είναι πρόταση. Ας αξιολογήσουμε αν αυτά που κάναμε ως τώρα ε, έχει νόημα να τα κρατήσουμε. Και όταν είπα ότι θυμάμαι την εποχή που δεν είχαμε αυτές τις αξίες, φυσικά εννοούσα την παρακολούθηση από το κράτος. Και από την αρχή που ασχολήθηκα με τα δημόσια, με τα κοινά, ε, αυτό ήταν το μέλημά μου. Και τώρα, πάλι στον κύριο ε, Λένερς από το ΕΛΚ. Για ένα λεπτό. ενδιαφέρουσα η συζήτηση για το δίκαιο και το EDPS, αν θα πρέπει να είναι ένας ουδέτερος νομικός εταίρος ή ένας πολιτικός εταίρος με συγκεκριμένες εκφράσεις πολιτικών επιλογών. Θα ήθελα λοιπόν να μου μιλήσετε για την διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αν θα αποτελέσετε έναν ουδέτερο παρατηρητή νομικό ή θα κάνετε πολιτικές παρεμβάσεις. Υπάρχουν και τα τεχνικά θέματα και τα νομικά. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων στον τομέα το νομικό και έλλειψη στον τομέα τον τεχνικό. Μόνο δύο έχετε προσλάβει. Έχετε πάρει μέτρα τον τελευταίο καιρό για να αντιμετωπίσετε το θέμα και τι θα κάνετε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την εύκολη ερώτηση την πρώτη αν πιστεύετε ότι το EDPS θα πρέπει να παίζει τον ρόλο του πολιτικού εταίρου. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν είναι ρόλος αυτός του EDPS να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Εμείς είμαστε εμπειρογνώμονες, εμείς μιλάμε για αξίες και δεν μιλάμε ε, για πολιτικές παρεμβάσεις δεξιά ή αριστερά δεν θεωρούμε ότι οι πολιτικές μας απόψεις πρέπει να μας συνοδεύουν στο γραφείο. Αυτό είναι κάτι το σαφές για τις δραστηριότητές μας, γιατί εμείς υποτίθεται ότι θα ελέγχουμε όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όταν προσπαθούμε να συμβουλέψουμε το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, ο ρόλος μας θα είναι να δώσουμε πρακτικές συμβουλές περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα μιλούσαν κυρίως οι δικηγόροι. Τώρα θέλουμε μια πολλαπλότητα γνώσεων στις υπηρεσίες. Ε, υπάρχουν πολλοί τεχνικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά και θα κατανοούν επίσης τις νέες λύσεις οι οποίες ε, θα ακολουθηθούν στο μέλλον όπως ε, ε, οι υπολογιστές Edge και άλλα μέσα. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να ακολουθήσουμε και να επενδύσουμε. Να δούμε ακριβώς τι είδους γνώσεις χρειαζόμαστε και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συνέργεια ανάμεσα σε μας και τις άλλες αρχές που έχουν ίσως εμπειρογνωμοσύνη σε άλλους τομείς. Τελευταία ερώτηση, Κλοντ Μωράες, ένα λεπτό. Να επανέλθω λίγο στο θέμα το οποίο έθεσε η κυρία Ιντβελτ Απαντήσατε σε βάθος σε πολλές ερωτήσεις. Το θέμα είναι ότι μπορείτε να μας δώσετε μια σωστή, ένα συμβουλευτικό κείμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάνετε νέες προτάσεις και τα λοιπά. Τελικά όμως, και για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, όταν υπάρχει ε, σε βάθος ε, αυξημένη και σωρία εμπειρογνωμοσύνης, περιπλέκονται τα πράγματα. Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα θέματα πάνω στα οποία δίδετε τις συμβουλές. Και δεύτερον για το θέμα του Cambridge Analytica. Βλέπετε ότι ε, οι πολίτες ε, βλέπουν ότι έχει γίνει κάτι λάθος και μας ρωτούν τι ακριβώς κάνετε για την πρόληψη αυτών των μεθόδων χρήσης των δεδομένων. Ε, τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να γίνει για να το θέσετε σαν προτεραιότητα. Κοιτάξτε, η καταχρηστική αν θέλετε παρουσία στο διαδίκτυο είναι κάτι το οποίο καλύπτεται και από το EDPS αλλά όχι στο σύνολό του. Ε, υπάρχει ένα τμήμα, αν θέλετε, ε, της Cambridge Analytica, της υπόθεσης, που έχει σχέση και με μας. Ε, η χρήση για πολιτικούς λόγους κάποιων δεδομένων είναι κάτι που υπάρχουν πολλές υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν, να τις κάνει να δραστηριοποιηθούν. Η ασφάλεια των δεδομένων, η οποία προκαλείται από τις πολιτικές δραστηριότητες, είναι επίσης κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και γι' αυτό θα πρέπει να πω ότι ένα από τα βασικά θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα ήταν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η χρήση των δεδομένων από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προετοιμασίες για τις ευρωεκλογές όπου τα δεδομένα δόθηκαν σε ε, υπηρεσίες επεξεργασίας εκτός των ευρωπαϊκών οργάνων. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά δεν μπόρεσε να λειτουργήσει σε επίπεδο ελεγκτικό και να ελέγξει εννοώ ακριβώς αυτά τα οποία περιλαμβάνονταν στις συμβάσεις που είχε κάνει. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά ζητήσαμε να τερματιστούν οι συμβάσεις αυτές και να διαγραφούν τα δεδομένα. Λοιπόν, βλέπω ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά, έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και το τελευταίο εξάμεινο είχα στο γραφείο μου έναν από τους βασικούς διερευνητές της υπόθεσης ε, Cambridge Analytica, ο οποίος ως εθνικός εμπειρογνώμονας συνεργάστηκε με μας. Σας ευχαριστώ κύριε Βεβερόφσκι για τη συνεργασία. Έχετε δύο λεπτά για μια τελική δήλωση αν θέλετε. Σας ευχαριστώ. Να θυμίσω κάτι το οποίο ήταν και στο γραπτό μέρος των απαντήσεών μας, στο θέμα της μαρτυρίας που έδωσα πριν έρθω σε αυτή την αίθουσα που ξεκινάει με ε, το πριν από 27 χρόνια όταν πρώτο μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οργανισμό που είχε ως ε, όραμα το δίκαιο κόσμο όπου υπάρχει σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ποικιλομορφία. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει ε, όθηση να κινούμε μέχρι σήμερα. Το κράτος δικαίου είναι η βάση των συζητήσεων μας, ε, η βάση είναι ο άνθρωπος, διότι δεν προστατεύουμε τα δεδομένα, προστατεύουμε τον άνθρωπο. Και η προστασία των δεδομένων δεν είναι παρά το εργαλείο για να πετύχουμε αυτό τον τελικό σκοπό. Ταυτόχρονα, να μην ξεχνάμε ότι διαφέρουμε ένας από τον άλλον. Υπάρχει πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη και είναι κάτι το οποίο αγαπάμε στο, σε αυτό το ευρωπαϊκό όραμα. Το γεγονός ότι μιλάμε τόσες γλώσσες, ότι συζητάμε τόσες κουλτούρες είναι μέρος αυτής της πρόκλησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να, αφήσω να ζω σε έναν κόσμο όπου αυτό το πρότυπο που έχουμε στην προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη αναγνωρίζεται ως κάτι το οποίο ε, είναι ένα πλεονέκτημα στην αγορά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα καινοτόμο τρόπο στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε τα θεσμικά όργανα που να ηγούνται με το, με το παράδειγμά τους ως e, ΕΦΙ δηλαδή μπορούν να, μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες για να κάνουν τα πράγματα καλύτερα από ό,τι έχουν γίνει μέχρι στιγμή. Αν έχουμε μια συζήτηση για το blockchain, ας μην συζητάμε απλά ποια είναι η πρόκληση που ε, αποτελεί, αλλά να θυμόμαστε και τα θετικά και τις επιτυχίες που θα μπορούσε να μας δώσει στη ψευδόνιμη χρήση των δεδομένων, που είναι κάτι που είναι κλειδί στον κανονισμό GDPR. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ όλα τα μέλη που επέβαλαν τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ για αυτό το δεύτερο γύρο ερωτήσεων και αποκρίσεων. Ευχαριστούμε κύριε Βιβυρόσκη, και για την παρουσίασή σας, τις προσπάθειές σας, τη ε, συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση και ε, εκτιμούμε την μακρά ε, σαδιοδρομία σας στον τομέα της προστασία των δεδομένων και το γεγονό ότι έχετε επιλεγεί σε αυτό τον μικρό κατάλογο. Συγχαρητήρια για τις προσπάθειες σας σε αυτό τον τομέα και καλή τύχη λοιπόν. Θα προχωρήσουμε με τον τρίτο υποψήφιο αυτής της βραδιάς σας. Ευχαριστώ. without further ado, it's late hour and we still have some time to go. So thank you for staying in the room this late hour. Σε ευχαριστώ που παραμένετε. Θα ακούσουμε τον τρίτο λοιπόν υποψήφιο. Επελέγεται ως τρίτος μετά από κλήρωση. Ε, σας καλωσορίζουμε παρόλα αυτά, ε, σας ε, συγχαίρομαι που έχετε επιλεγεί ανάμεσα στους τρεις. Συνειδητοποιούμε ότι έχετε διανύμει το κουρούκουλουμ σας. Ακολουθούμε μία συγκεκριμένη μέθοδο. Έχετε πέντε λεπτά για την παρουσίασή σας και μετά θα ακολουθήσουν 10 ερωτήσεις, ενός λεπτού η κάθε μία και δύο λεπτά η απάντησή σας για κάθε ερώτηση και μετά έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πάντοβα, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι που μου δώσατε ε, τόσο αργά την δυνατότητα να σας παρουσιάσω τις απόψε μου. Θέλω να συγχαρώ τον Τζοβάνι Μπουταρέλη με τον οποίο έχω συνεργαστεί ε, επανειλημμένα. Στον τομέα της προστασίας των δεδομένων έχω κάνει μία περιστροφή 360 μοιρών. Ήμουν υπάλληλο ανώτατος στην Γενική Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ήμουν ε, υπεύθυνο της ρυθμιστικής αρχής, της ΚΝΙΛ, που είναι η υπηρεσία που ασχολείται με την προστασία των δεδομένων και ήμουν και επίτροπος στον τομέα της ενέργειας και τον smart meter και των smart ε, ε, δικτύων. Έχω δημοσιεύσει άρθρα σε πάρα πολλά διεθνή περιοδικά. Είμαι στρατηγικός ε, σύμβουλος της Αγγλικής Ρυθμιστικής Αρχής. Ασχολούμαι με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ε, προστασίας ε, των δικαιωμάτων του πολίτη. Αυτή η επισκόπηση μου δίνει τη δυνατότητα να γεφυρώνω τα, δίκαια με την, τα δικαιώματα με την τεχνολογία, τα δικαιώματα με το δίκαιο. Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η ανεξαρτησία. Όταν έχω οργανώσει ε, το πρώτο έλεγχο φακέλου των αστυνομικών δεδομένων στη χώρα μου, ε, εν πλήρη ανεξαρτησία και στα πλαίσια της δραστηριότητας της ΚΝΙΛ και επίσης ε, έχω εργαστεί ως υπερασπιστής προμπόνου. Ε, το μάλιστα αυτό με οδήγησε και στο Κορεπέρ πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχουν ανησυχίες από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών ε, νιώθουν ότι, ελέγχουν, ότι δεν ελέγχουν μάλλον τα δεδομένα τους. Η προστασία των δεδομένων τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει πολύ. Ένα θέμα κάποτε για ειδικού έχει γίνει κεντρικό για πολλούς. Είναι κεντρικό γιατί επηρεάζει και άλλες ε, ε, θεμελιώδεις ελευθερίες, ελευθερία διακίνησης ανώμημα, Έχετε επίσης και εκλογές οι οποίες μπορεί να παραποιηθούν και αναφέρομαι εδώ στο Cambridge Analytica. Μπροστά σε αυτές τις ανησυχίες δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Να ενισχύσουμε τα κοινοβούλια, ε, έτσι θα προστατεύσουμε τις αξίες μας σαν Ευρωπαίοι και θα πρέπει επίσης να μετατρέψουμε και τον ρόλο, να αλλάξουμε τον ρόλο του ελεγκτή. Το business as usual δεν είναι μια επιλογή. Θα συνεχίσω τα αγγλικά στα πλαίσια των τεσσάρων μέτρων που θέλω να λάβω για να βελτιώσω τη λειτουργία της υπηρεσίας. Λοιπόν, πολυεπιστημονικότητα ή διεπιστημονικότητα, αύξηση δραστηριοτήτων, έλεγχος, να μου επιτρέψετε βέβαια να είμαι λίγο πιο αναλυτικός, διεπιστημονικότητα, περισσότερη ε, μηχανική στον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης. Ε, χρειάζεται να έχουμε σωστές συμβουλές σε τεχνολογικό επίπεδο. Full activity. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αρκούμεθα ε, στις εθνικές συμβουλές, αλλά θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με όλους, λαμβάνοντας επόψη και την εξάρτηση την οποία μπορούμε να έχουμε από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σαν παράδειγμα η Κίνα και θα πρέπει επίσης να είμαστε διαθέσιμοι για να σας δίνουμε συμβουλές όποτε το επιθυμείτε. Και τέλος, θα πρέπει να είμαστε ο ελεγκτής ο οποίος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι σαφές λοιπόν ότι απαιτείται επαϊοσύνη, ανεξαρτησία και γνώση. Νομίζω ότι είμαι ένας πραγματικός Ευρωπαίος, αναγνωρίζω τις αξίες μας, έχω και γαλλικές εμπειρίες, έχω επίσης και ιταλική ε, προέλευση και το λέει το όνομα ε, της, ε, της οικογένειάς μου. Είμαι και γιος Σουηδής και γνωρίζω και τη Σουηδική. Ευχαριστούμε κύριε Να Είστε σίγουρος ότι έχετε τον σεβασμό όλης της Επιτροπής που ήσασταν και τόσο σύντομα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Η κυρία Μετσόλα από το ΕΛΚ για ένα λεπτό έχει την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Παντοβά για την παρουσίασή σας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το επόμενο μέτωπο σε επίπεδο δεδομένων και θα απαιτηθούν τεράστιες διαδικασίες επεξεργασίας. Θέτει αυτό πολλά ηθικά ζητήματα. Ποιον ρόλο βλέπετε ότι θα έχει ο Ευρωπαϊκός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ε, για να καταστήσει δυνατό ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει ενωμένη. Πώς θα υπάρχει προστασία και καινοτομία ταυτόχρονα και πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών θα προστατεύουν προστατεύονται, ειδικά όταν έχουμε συνεργασία με μη Ευρωπαίους ε, παίχτες. Ε, γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιοι που προτείνουν ε, δικαιώματα ιδιοκτησίας. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Μετσόλα. Έχετε το λόγο κύριε Παντοβά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ευρωβουλευτά. Όντω η τεχνητή νοημοσύνη είναι το νέο μέτωπο. Αναφέρατε όγκο, ε, νούμερα. Είμαστε σε τεράστιους όγκους δεδομένων αυτή τη στιγμή, 85% αυτών δεν χρησιμοποιούνται από τις εταιρείε. Doctate ονομάζονται αυτά. Ταυτόχρονα όμως συγκεντρώνονται σε κάποιους συγκεκριμένους operators. Έχουμε λοιπόν τη διάχυση και την συγκέντρωση και οι τομείς αυτοί δεν είναι έτσι λοιπόν είμαστε λίγο στριμωγμένοι μεταξύ δύο μοντέλων. Έχουμε το αμερικάνικο μοντέλο, δεν υπάρχει μια γενικότερη νομοθεσία όπως το GDPR, υπάρχει μόνο τομεακή νομοθεσία ή ένας ε, δικαστής που επεμβαίνει και μετά υπάρχει και το μοντέλο της Κίνας με συλλογή τεράστια συλλογή δεδομένων και παρεμβάσεις. Εμείς νομίζω ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν ανθρωπινό, ανθρωπιστικό και σωστό τρόπο ε, χρήσης και συλλογής δεδομένων. Με λογοδοσία. Ε, η Κομισιόν πρότεινε ότι θα το κάνει σε 100 μέρες. Ο ευρωπαϊκός τρόπος είναι η αξιόπιστη χρήση της Τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν εμπιστευόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, θα χάσουμε την πίστη στη δημοκρατία, στη μας και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Άρα, έχουμε το πλεονέκτημα στην Ευρώπη ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε μια μορφή νομοθεσία στο GDPR. Υπάρχουν πολλές διατάξεις που λένε, για παράδειγμα, ότι δεν χρειάζεται να είσαι το αντικείμενο μιας απόφασης για να ε, ε, υπόκεισε σε επεξεργασία δεδομένων. Υπάρχουν όμως και κενά στο GDPR. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάτι για να πληρώσουμε αυτά τα κενά. Ας πούμε η διαφάνεια του αλγορίθμου, η ορατότητα. Ο ρόλος του EDPS είναι να βοηθήσει στη δημιουργία αυτών των νέων κανόνων και να μην έχουμε έτσι πειραματισμούς όπως το Sandbox ε, στο ICO. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Δύο ε, λεπτά για κάθε απάντηση. Α, βλέπω τώρα το χρονοδιακόπτη. Ναι, εκείνη για να το θυμάστε. Ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση. Δεύτερη, η κυρία Σίπελ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι σε αυτό το μεγάλο ερώτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Και εσείς μεταξύ άλλων μιλήσατε για τη διαφάνεια και τη σημασία του GDPR. Όμως, μπορείτε να μας πείτε ποια θα είναι κάποια καλά παραδείγματα διασφάλισης της διαφάνειας, όχι μόνο για τις αρχές αλλά και για τους πολίτες. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι από μόνη της θα εξελίσσεται. Τι είδους έλεγχο θα μπορούμε να έχουμε. Χρειαζόμαστε επιπλέον μέτρα από το GDPR για να το διασφαλίσουμε. Θα επανέλθω και στις γραπτές απαντήσεις σας. Υπογραμμίσατε γενικά τη σημασία της ανεξαρτησίας από τη δική σας άποψη λοιπόν και πλευρά. Ποιος είναι ο ρόλος του EDPS ε, και του Συμβουλίου ο επόπτης και το Συμβούλιο είναι αρκετά ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή ή πρέπει να ενισχυθούν για να έχουν ακόμα περισσότερη ανεξαρτησία στην εργασία τους. Κύριε Παντοβά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, δύο ερωτήσεις στην ερώτησή σας. Αν χρειαζόμαστε επιπλέον μέτρα για να ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και το είπα και πριν, στην, ως απάντηση στην κυρία Μετζόλα, ναι είναι η απάντηση. Το GDPR δεν καλύπτει όλα τα θέματα της τεχνητής νομιμοσύνης. Productability, redressability, πώς ε, μετράς ε, την, ε, τις διακρίσεις αυτό νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί στους κανονισμούς μας, να έχουμε καλύτερα μέτρα διαφάνειας και επεξηγηματικά μέτρα, είτε με κώδικες δεοντολογίας, είτε και με άλλο τρόπο. Ε, π.χ. να έχει ο ρυθμιστής κάποιους πόρους IT ε, στη διάθεσή του. Βέβαια, δεν μπορείς να είσαι ανεξάρτητος αν έχεις μόνο νομικά μέτρα και όχι τεχνολογικά. Δεν θα κατανοείς τον κόσμο που ζεις, ούτε την τεχνολογία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε διάφορα είδη, διάφορες ειδικότητε, π.χ. μηχανικούς, ε, που θα μας δίνουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, γιατί αλλιώς ε, δεν θα αντιμετωπίσεις την πρόκληση. Όταν ήμουν ε, ε, στην ΚΝΙΛ ε, είχα επί τρία πολλαπλασιάσει τον αριθμό των μηχανικών. Έτσι είχαμε το στάνταρ της τεχνολογίας που θέλουμε να έχουμε ως συμβούλους για το GDPR. Άρα δεν είναι μόνο θέμα πόρων, αλλά και κατανόησης του τι σημαίνει και δυνατότητας να δώσεις ε, σωστή και, μια σόφρονα συμβουλή. Εγώ είμαι δικηγόρος. Ξέρω ότι δεν είμαι τέλειος σε όλα και ότι υπάρχουν οι πληροφορικάροι που μπορούν να με βοηθήσουν. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Φέλτα από το Ρηνιού. Ευχαριστώ κύριε Πάντοπα για την εισαγωγή σας. Τρεις γρήγορες ερωτήσεις. Πρώτον, υπάρχουν Υπάρχουν πολλές προσδοκίες από το EDPS, το νομικές και τεχνικές. Αυτό που λείπει είναι το σθένος, η δύναμη, διότι ε, παραβλέπονται εντελώς οι γνώμες της, από την Κομισιόν. Τι θα δω, πώς θα δώσετε περισσότερο, περισσότερη ισχύ στο EDPS και πώς θα ενισχύσετε την επιβολή. Η Επιτροπή Εμπορίου τον ΗΠΑ έχει επιβάλει, για παράδειγμα, πρόσημο 5 δις στο Facebook ε, και τα πρόστιμα που παίρνουν στην Ευρώπη είναι για γέλια. Ε, και πώς θα ενισχύσετε λοιπόν την επιβολή. Επίσης, στο θέμα της διαφάνειας θέλω να ε, δω. Ε, έχω ζητήσει από το EDPB να δημοσιεύσει τα πρακτικά της. Εσείς θα στηρίζατε αυτή την έκκληση που έχω κάνει. Κύριε Πάντοβα, για δύο λεπτά. Τρεις ερωτήσεις σε δύο λεπτά. Ε, μερικά δευτερόλεπτα για κάθε απάντηση. Η αξιολόγησή σα είναι ότι οι γνώμες ε, του EDPS παραβλέπονται από την Κομισιόν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και η δέσμευσή μου είναι να, για να βελτιώσουμε την κατάσταση είναι πρώτα απ' όλα να δουλεύουμε από τα πρώτα-πρώτα στάδια όσο πιο νωρί μπορούμε έτσι ώστε να έχουμε κάποια επιρροή και να διασφαλίζουμε συνέπεια ανάμεσα στις διάφορες πρωτοβουλίες, ε, διότι υπάρχουν κάποια σιλό και σε επίπεδο της Κομισιόν και δεν γνωρίζουν πάντα και τι συμβαίνει αλλού. Δεύτερο, αν δεν είστε ικανοποιημένοι, μπορεί να χρησιμοποιείτε τα δημόσια μίντια. Μπορείτε ε, να δημοσιοποιείτε κάποια θέματα. Ε, θα πρέπει να είστε επιλεκτικός για να είστε αποτελεσματικοί αλλά μπορείτε να ε, το ζητήσετε δημόσιο. Τρίτη επιλογή, ε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα, αλλά όπως είπα, θα πρέπει να επιλέγει την υπόθεση. Δεν μπορεί να το κάνει για κάθε υπόθεση. Πρέπει να είσαι επιλεκτικός, διότι μπορεί να χάσει πολλά. Τώρα, για την επιλογή, ε, επιβολή. Το EDPS δεν είναι εθνικό ρυθμιστή. Έχει μικρή δύναμη σε ό,τι αφορά τι κυρώσει. δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ε, επιβάλλουμε. Υπάρχει χώρος βελτίωσης στον τομέα της επιβολής. Στις γραπτές απαντήσεις είπα ότι θα διοριστώ. Θα δημοσιεύσω ένα πρόγραμμα ετήσιων ε, επιθεωρήσεων και θα λογοδοτούμε. Ε, με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε την περιοχή μας. Λέμε τι θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε αυτά που λένε. Με. Ε, σχετικά με τη διαφάνεια ε, και αυτό ε, αφορά την ελευθερία πληροφόρησης, και ενημέρωσης θα στήριζα αυτό το αίτημα, δεδομένου ότι είναι μέσα στα όρια του νόμου φυσικά. Ευχαριστώ. Η πράσινη, κύριε Μπρέιρ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πάτοβα. Είχαμε την χαρά να συναντηθούμε πρόσφατα και να συζητήσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις ε, του επόπτη προστασίας δεδομένων και αν θυμάμαι καλά είπατε ότι σας αρέσει η προσέγγιση της Βρετανικής ICO, της Επιτροπής ε, για την Εποπτεία της Προστασίας των Δεδομένων ε, σε σύγκριση με άλλες αρχές που τείνουν να κάνουν σαφείς δηλώσεις και άκαπτες δηλώσεις και αποφάσεις, ενώ η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου, είπατε, είναι πιο συνεργατική και χρησιμοποιούνται οι... Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ακριβώς ποια είναι η ιδέα σας ε, σε αυτό. Και δεύτερον, Ποια είναι η άποψή σας ε, ε, στην, ε, στις νόμους υποχρεωτικής κράτησης δεδομένων. Απάντηση από τον κύριο Πάτοβα. Ευχαριστώ, όπω είπατε κύριε ε, Βουλευτή. Είμαι στρατηγικός σύμβουλο της ICO για το θέμα του sandbox, των δοκιμαστηρίων δεδομένων και την προστασία δεδομένων. Είναι ε, ενδιαφέρον, αλλά ε, ε, λειτουργεί ως καλός ρυθμιστής. Δεν δίνει μόνο συμβουλές, αλλά είναι και δυνατός στην επιβολή. Έχει σαφή στρατηγική, γιατί το ψηλότερο πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προέρθει από το ICO. Το ICO έχει πραγματιστική προσέγγιση και πολύ λογική σε συνεργασία με όλους τους συμμετόχους, με δημόσια διαβούλευση, έχει ε, δίνει στήριξη, παρέχει εργαλεία, ε, αλλά από την άλλη πλευρά είναι δυνατός ε, οργανισμός στην επιβολή και ότι αν υπάρχει αυτή η ισορροπία, την οποία θα υποστήριζα και εγώ, είναι δίκαιη και ε, ισορροπημένη η προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική κράτηση δεδομένων, ε, ήμουν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπέρ αυτής της υπόθεσης. Είναι η υπόθεση που στηρίζεται στην Οδηγία 2258 και ε, για την κράτηση, υποχρεωτική κράτηση των δεδομένων, μια νομολογία που έχει θεσπιστεί για πολλά χρόνια τώρα και Πιστεύω ότι στο θέμα της υποχρεωτικής κράτησης θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στις υποθέσεις που θα το επέτρεπαν αυτό και να έχουμε τα ένδικα μέσα και την διαφάνεια. Αλλά ήμουν εναντίον ε, στο γαλλικό δίκαιο να μην υπάρχει, ότι δεν, να μην υπάρχει υποχρεωτική απόφαση ε, σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Είναι απλά γνωμοδότηση μιας ανεξάρτητης αρχής που δεν επαρκεί και δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα στοιχεία. Θα ήθελα να σας πω περισσότερα, ε, διότι αγόρευσα για 15 λεπτά στο θέμα αυτό. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ. Τώρα, κύριος Καρό, για ένα λεπτό έχετε το, το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πάντοβα. Έχουν τεθεί πολλές ερωτήσεις σχετικές με τον ρόλο του influencer της ε, συγκεκριμένης υπηρεσίας. Είδα στο curriculum Βίτε σας κάποια στοιχεία που δεν είδα στους άλλους υποψήφιους. Ε, έχετε κάνει πολλές δημοσιεύσεις τα αγγλικά σε συγκεκριμένα περιοδικά όπως το Oxford International of Comparative Law και στο Columbia Law Review. Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες και από ό,τι καταλαβαίνω, ελπίζω να μην κάνω λάθος, χρησιμοποιήθηκαν και για αποφάσεις που πήρε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το δικαίωμα εξάλληψης της μνήμης, αν θέλετε. Το θέμα λοιπόν είναι αν αυτή η δραστηριότητα η ερευνητική είναι σημαντική για σας και αν συνεχίσετε ε, ε, τον ρόλο αυτό και αύριο. Απαντήστε κύριε Παντοβά. Θα απαντήσω στα γαλλικά γιατί η ερώτηση είναι γαλλική. Ε, εδώ και 15 χρόνια έχω μια συνεχή ερευνητική δραστηριότητα και σε πρακτικό επίπεδο, είτε ως ρυθμιστής είτε ως δικηγόρος, χρειάζομαι ε, κάποια απόσταση και ακριβώς η διδασκαλία και η έρευνα με βοηθά. Τρία είναι τα θέματα. Εδαφική κάλυψη του δικαιωμάτων των δεδομένων, ιδιοκτησία των δεδομένων και ο σύνδεσμος ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων και την καινοτομία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο και σε επίπεδο πρακτικής ε, το άρθρο που συνυπογράφω με τον καθηγητή Βίκτορ Σόνμπεργκερ που είναι καθηγητής στην Οξφόρδη ασχολείται με το πώς αυτά που λέγαμε big data, τώρα λέμε τεχνητή νοημοσύνη, συνδέεται ε, και είναι συμβατή με τις αρχές της υπηρεσίας μας και τι πρέπει να γίνει για να είναι συμβατά όλα αυτά. Αυτό είναι ρόλος ενός ρυθμιστή. Όπως είπατε είναι στον τομέα του influencer. Ένας ρυθμιστής θα πρέπει να διαδίδει μέσα από συγκεκριμένες σκέψεις, μέσα από συγκεκριμένη αρχιτεκτονική των γνώσεων. Αλλά εγώ συνδυάζω αυτό και με την πρακτική. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί ο supervisor ε, δείχνει επίσης ε, και το τι κάνει η Ένωση προς τα έξω. Έχει και ρόλο πρέσβη θα έλεγα και θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει την αυτόνομη σκέψη η οποία μπορεί ε, να βοηθήσει και το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, στο δικαίωμα δηλαδή στη διαγραφή των στοιχείων και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό λοιπόν η έρευνα με βοηθά να δίδω σωστές συμβουλές στους νομοθέτες. Η Σιάρη, κυρία Κάνκο. Ευχαριστώ κύριε Παντοβά. Με χαρά διαπιστώνω ακριβώς την επιθυμία που έχετε να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις και τις αλλαγές της τεχνολογίας τις οποίες δεν προλαβαίνουν οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. <clears throat> το digital sovereignty είναι κάτι το οποίο συζητιέται συνεχώς. Αν θέλουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε μια συγκεκριμένη ασφαλή διαχείριση σε συνεργασία με τους φίλους μας, τους δημοκράτες ενώ στον υπόλοιπο κόσμο, μπορούμε να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και την παρανομία και να κρατήσουμε το διαδίκτυο ασφαλές μόνο μέσω της συνεργασίας. Ένα παγκόσμιο πλαίσιο προστασίας προτάθηκε από τους Ιάπωνες στο G20 στις αρχές του 19. Μπορούμε να το πετύχουμε στο εγγύς μέλλον. Είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Είναι ρεαλιστικό. Ο κύριος Παντοβά δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Το ερώτημα του να υπάρξει ένα παγκόσμιο πλαίσιο είναι ένα ερώτημα το οποίο συζητάμε οι ειδικοί της προστασίας των δεδομένων εδώ και 30 χρόνια. Η Ευρώπη ήταν πράγματι η πρώτη ήπειρος η οποία επεξεργάστηκε αυτού του είδους το πλαίσιο με την αρχική σύμβαση, με την οδηγία του 95 και με την αρχή της συγκεκριμένη σήμερα. Πίσω από το νομικό πλαίσιο υπάρχουν κάποιες αξίες θεμελιώδεις βαθύτατα ευρωπαϊκές. Υπάρχουν ε, άρθρα που καλύπτονται και από τη χάρτα για τα δικαιώματα και δεν είναι εύκολο να προωθήσει κανείς ένα επίπεδο προστασίας που να εδράζεται στις ίδιες αξίες. ανάμεσα στις ε, δύο ε, ακτές του Ατλαντικού. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες συγκλήσεις, αλλά υπάρχουν και διαφορές σε σχέση με την έννοια της ιδιωτικότητας. Κάποιες χώρες μάλιστα όπως η Κίνα έχουν μια ολιστική αντίληψη κάτι το, για την κοινωνία, κάτι το οποίο σε επίπεδο ουμανιστικό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Είναι εδώ και πολύ καιρό λοιπόν, από το 2008 στη διάσκεψη της Μαδρίτης έγινε συζήτηση για διεθνή στάνταρ στην προστασία των δεδομένων. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο αλλά απαιτείται χρόνος για να το πετύχουμε. Και δεν θα έχουμε μάλλον τους ίδιους μηχανισμούς γιατί δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα ελέγχου πρέπει να κάνουμε διάλογο με τις διαφορετικές χώρες, αλλά δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε συνταγές. Έχουμε ένα ηγετικό ρόλο, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αλαζόνες. Ο κύριος Αρένα για την ΚΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πρόσφατα ε, κάποιες αποφάσεις για την αύξηση Τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων για θέματα ασφαλείας. Θα υπάρξουν και νέες πρωτοβουλίες ε, στον τομέα της διαλειτουργικότητας των μεγάλων δεδομένων, βάσεων δεδομένων, για τη δικαιοσύνη, ε, για το PNR και τα λοιπά. Αν και καταλαβαίνω ότι η απάντηση μπορεί να είναι λίγο περίπλοκη, πώς εσείς θεωρείτε τη σημερινή κατάσταση δικαίωμα στην ιδιωτικότητα σε συνδυασμό με τα μέτρα παρακολούθησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πώς τα πού οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορέσει η Ένωση να επηρεάσει και τους Αμερικανούς νομοθέτες. Ευχαριστώ. Είναι θέμα που άπτεται και της πολιτικής στον τομέα αυτό. Να πω ότι ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν είχε πει ότι μπορεί να θυσ... αν κάποιος θέλει να θυσιάσει τις ελευθερίες του υπέρ της ασφάλειας θα χάσει και τα δύο. Συνεπώς λοιπόν ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές επιθέσεις και απειλές και υπάρχει ανάγκη για ισχυρή συλλογή δεδομένων και κοινή διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά όχι εις βάρος των δικαιωμάτων αυτό είναι κάτι το οποίο είχα πει και στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο λέγοντας πως αν δεν γνωρίζει κανείς ότι είσαι υπό επίβλεψη, πώς θα αναζητήσεις τα δεδομένα τα οποία σε αφορούν. Είναι επίσης αλήθεια ότι αν είσαι ενήμερος, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην συνεχίσει η παρακολούθησή σου ή ο έλεγχός σου και στα πλαίσια των νομικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην Γαλλία, σαν παράδειγμα, στον τομέα αυτό δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ε, των υποκείμενων σε έρευνα. Συνεπώς λοιπόν πράγματι θέλει προσοχή και από τις δύο πλευρές γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε και τους δύο. Έχει το λόγο η κυρία Φόξ. Κύριε Παντοβά, ε, συμφωνά για την έρευνα και τους ε, μηχανικούς πληροφορικής, όμως ε, για την πολιτική καμιά φορά η αξία της ελεύθερης γνώμης είναι πιο σημαντική από την προστασία των δεδομένων. Άρα δεν ξέρω αν αυτό είναι για να βρούμε ένα νέο τρίκ για να σταματήσει το δικαίωμα στον ελεύθερο λόγο. Καλό θα είναι λοιπόν ε, να επιτρέπεται στα άτομα να ε, διαγράφονται τα δεδομένα τους. Τώρα τι γίνεται όταν απαιτούν ε, αυτά που λένε στο facebook να διαγράφονται και μετά πέφτουν στα χέρια του δικαστηρίου. Νομίζω ότι φτιάχνεται ένα τεράστιο φάργολ γύρω από την Ευρώπη Παρόμοιο με αυτό της Κίνας ε, που λέει ποιος θα έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και ζητά τα πάντα. Ε, θα ήθελα λοιπόν εάν ο Ευρωπαίος Επόπτης θα δίνει ε, στα άτομα τη δυνατότητα να μιλούν ελεύθερα και να διατηρούν τα δεδομένα τους ή όχι. Ah, <laughs> Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι η συζήτηση της επικράτειας ε, στην οποία έχουμε δικαιοδοσία έχει, έχει μεγάλη σημασία και υπάρχει και το δικαίωμα του ελεύθερου λόγου και της πρόσβασης στα δεδομένα σου. Έτσι λοιπόν ε, το θέμα αυτό ε, της επικράτειας ήταν πολύ σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί αν πας πέρα από την επικράτειά σου θα πρέπει να έχεις και αντίμετρα από άλλα κράτη, τα οποία θα, θα επιτρέπουν στους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Το να έχεις λοιπόν ένα πολύ ευρύ και καθολικό πεδίο από ευρωπαϊκή άποψη θα ήταν ένα μειονέκτημα ε, καθώς θα είχαμε κάποιες χώρες λιγότερα δημοκρατικές που δεν θα μας έδιναν πρόσβαση σε δεδομένα. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Δικαστήριο βρήκε λοιπόν τη σωστή ισορροπία μεταξύ στην πρόσβαση στα δεδομένα και στο δικαίωμα της λύθης, γιατί πραγματικά όταν ε, μιλάμε για λύθη δεν ε, διαγράφονται τα δεδομένα, απλά βγαίνουν από τις μηχανές αναζήτησης. Όταν γίνεται αυτό, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να γίνεται στο πεδίο της ευρωπαϊκής επικράτειας βάσω ε, ε γεωτοποθέτησης για να μην μπει σε κίνδυνο η πρόσβαση των πληροφοριών από ε, την πλευρά των Ευρωπαίων πολιτών και να μην υπάρχουν και αντίπεινα από τις άλλες χώρες. Αυτό ακριβώς ήταν και οι μελέτες μου και τα άρθρα μου. Η διατήρηση του δικαιώματος ε, στον ελεύθερο λόγο και στην πρόσβαση στα δεδομένα έχοντας όμως και μια ισορροπία μεταξύ αυτού και ε, μεταξύ ε, των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κοινό Λέναρς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πάνοβα. Συζητήσαμε και με τους άλλους ε, υποψήφιους τον ε, ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας. Αν θα πρέπει να είναι ένας αδέκαστος πολιτικός ε, δράστης ή να είναι ένας άνθρωπος με, πολιτική, με πολιτικό όραμα και πολιτική δράση. Πώς βλέπετε εσείς τον επόπτη και το ρόλο του λοιπόν. Δεύτερον, έχετε δουλέψει με τους θα δουλεύετε μάλλον με τους Ευρωπαίους εθνικούς επόπτες. Πώς αξιολογείτε αυτή τη στιγμή τις εθνικές αρχές και τους επόπτες. Ε, υπάρχουν εκατομμύρια δεδομένα πολιτών που αποθηκεύονται αυτή τη στιγμή σε κάποια μόνο κράτη-μέλη. Πώς θα βοηθήσετε, για παράδειγμα, τα μέλη ως ε, ευρωπαίσωπο από τις προστασίες δεδομένων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, νομίζω ότι για να είσαι αδέκαστος πρέπει να έχεις λάβει πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το ρόλο. Έχω εκπαιδευτεί γι' αυτό, ήμουν στο κογκρέσο της, στη Γαλλία και εκεί το να είσαι άδεκαστος ήταν θέμα επιβίωσης, γιατί το να παίρνει θέση κάθε πέντε χρόνια που θα άλλαζε κυβέρνηση θα σήμαινε ότι θα είχες μεγάλο πρόβλημα. Δεκαπέντε χρόνια ήμουν εκεί. Το να είσαι όμως αδέκαστος ως ρυθμιστής δεν σημαίνει ότι δεν λες αυτό που πιστεύεις αλλά ούτε και σημαίνει ότι μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι. Δίνεις καθοδήγηση, λες ε, τις συμβουλές σου και φυσικά μετράς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, αλλά δεν παίρνεις εσύ το ρόλο του νομοθέτη, είσαι ο, συμβουλε, ο σύμβουλος. Είσαι αμερόληπτος και αυτό αρκεί. Δεν θα πρέπει να γίνεις κάτι παραπάνω από σύμβουλος, δηλαδή δάσκαλος ή καθηγητής. Τώρα για το ρόλο των εθνικών αρχών, για τους εθνικούς επόπτες, ξέρω ότι γενικά δεν υπάρχουν πόροι και το GDPR έχει αυξήσει το βάρος. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Η μεγαλύτερη είναι το SEO που έχει 600 άτομα και ακόμα αντιμετωπίζει προβλήματα σε επίπεδο προσωπικού αλλά και δεξιοτήτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μηχανικός πληροφορικής ε, και οικονομολόγους. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Η Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, τους έχει αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και σε κάποια ε, κρατήδια στη Γερμανία και σε κρατικό επίπεδο στη Γαλλία. Ίσως λοιπόν η βελτίωση θα ήταν ένα δίκτυο που θα συλλέγει τους πόρους και θα ανταλλάσσει εμπειρογνωμοσύνη στον τεχνολογικό τομέα. Ζητώ συγγνώμη, μπερδεύω τη γλώσσα είναι λίγο αργά. Ο κύριος Μωράς για την τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια επανάληψη στις ερωτήσεις, αναπόφευκτα αυτή είναι η τελευταία. Επανέρχομαι στην προσέγγισή σας. Σας ρώτησαν για το ICO και για το γεγονός ότι ήσασταν Σύμβουλο ε, και δίνατε συμβουλέ στην Κομισιόν. Η Κομισιόν λοιπόν, ας πούμε ότι φτιάχνει μια νέα πρόταση, εσείς δίνετε τη συμβουλή σας ε, και σας αγνοούν. Πώς θα προσεγγίσετε αυτή την κατάσταση, γιατί αυτό το θέμα είναι μεγάλο για τον Ευρωπαίο ότι πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο, την κατεύθυνση τέλο πάντων και την νομοθεσία. Πώς θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση, πώς θα περάσετε τη γνώμη σας. Και υπάρχει και το θέμα του Cambridge Analytica. Στο μυαλό των ανθρώπων ακόμα υπάρχει παρέμβαση στις εκλογές και συνεχίζονται να πολλαπλασιάζονται αυτές οι μέθοδοι, οι μεθοδολογίες. Πώς ε, θα περάσετε στην, στο κοινό ε, την ε, δική σας άποψη για το πώς θα λύσουμε αυτό το θέμα. Παρακαλώ, η τελευταία σας απάντηση. Ναι, κατανοώ αυτό που λέτε ότι κάπο, πολλές, πάντοτε αγνοούν τις συμβουλές μας και υπάρχει ματέωση από ε, λόγω αυτού. Έτσι είναι τα πράγματα σύστημα σήμερα και δεν ξέρω αν θα το αλλάξω εγώ. Όταν σε αγνοήσουν έχεις πολλές επιλογές. Ίσως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να παρέμβεις στα πρώτα στάδια όταν έχουμε το σχέδιο κανονισμού. Ξέρω από προσωπική εμπειρία ότι αν πας πολύ αργά να παρέμβεις, όλες οι σημαντικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Αν θέλεις πραγματικά να έχεις κατάσταση win-win, με την Επιτροπή θα πρέπει να παρέμβεις στο πιο πρώιμο στάδιο στο σχέδιο, ούτε καν στο σχέδιο. Πιο πριν, όταν υπάρχει η άτυπη ανταλλαγή απόψε. Αυτό όμως ε, που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ποτέ 100% δεν λαμβάνονται υπόψη συμβουλές. Υπάρχει αυτή η απογοήτευση, είναι πολλές φορές φάσεις πολιτικές, η Κομισιόν δεν θέλει να πάρει συγκεκριμένη θέση. Εσύ δεν είσαι ο νομοθέτης και όταν έχουμε πολύ σοβαρά περιστατικά, όπως είπα πριν και στην κυρία Ινβέλτ, μπορείς να βγεις δημοσίως. Όταν είσαι μικρή αρχή, καλό είναι όταν έχεις μια καλή ιστορία να πεις, να τη βγάλεις στη δημοσιότητα και τέλος θα ακουστείς. Ξέρω ότι παίρνει χρόνο, ε, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ίσως ακόμη πρέπει να πας και στο δικαστήριο. Βέβαια, αν είσαι προμηθής, αν τα κάνεις όλα σε πρώιμο στάδιο και έχεις τα δικαστήρια ως τελευταία λύση, συν το χρόνο θα κερδίσεις σε επίπεδο επιρροής. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλα τα μέλη για την ε, υπομονή σας που ήσασταν εδώ, που μας ε, δώσατε τη δυνατότητα αυτή αυτές ε, οι ακροάσεις, η έκτακτη αυτή συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ, να έχει τόσο καλό περιεχόμενο. Ήρθαμε εδώ για ένα πολύ καλό λόγο. Είχαμε αυτούς τους τρεις ε, εξαιρετικούς υποψήφιους. Συγχαρήκαμε τους δύο προηγούμενους και συγχαίρουμε και εσάς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ήσασταν εδώ. Παρακαλώ, θέλατε να πείτε κάτι άλλο? Όχι? Ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Πήγα λίγο στην Ολομέλεια, αλλά να γύρισα. Ήθελα να πω ότι εκτιμούμε το ότι ήσασταν ο τελευταίο, ότι ήσασταν κι εσείς από τους πολύ σημαντικού ε, υποψήφους, αλλά έχετε δύο λεπτά για να κάνετε την τελευταία σας ε, δήλωση. Απολαύστε τα. Ευχαριστώ καταρχάς που μου δώσατε τη δυνατότητα να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Έχω μόνο δύο λεπτά. Θα θέλαμε ώρες να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Όμως θα αναφερθώ στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να καθησυχάσουμε και να μείνουμε με τα σκαρπούς του παρελθόντος. Ε, πρέπει να βρούμε νέες μεθόδους. Η αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων είναι σημαντικό στοιχείο, γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε εμά, δεν υπάρχει ούτε στην προστασία δεδομένων, ούτε οι πολίτες μας αισθάνονται ασφαλείς, γιατί δεν εμπιστεύονται τους παρόχους και τις υπηρεσίες. Γι' αυτό χρειάζομαστε κάποιον που είναι ανεξάρτητος και ανοιχτό σε διάλογο. Νομίζω ότι αυτό το κατέδειξα. Θέλουμε κάποιον που να κοιτάει στο μέλλον, να φτιάχνει γέφυρες και όχι τείχους, όπως ε, πιστεύω ότι είμαι και κάποιον ο οποίος είναι ε, στεναρός και απόλυτος όταν ε, χρειάζεται. Έχω εμπειρία και σε ιδιωτική εταιρεία και στο δημόσιο και ξέρω πολύ καλά ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό, οπότε ψηφίστε μαύρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. so much. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάντοβα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, για τη δήλωσή σας. Σας χαίρομαι που φτάσατε στο τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας ε, στην Επιτροπή μας. Ε, ε, η διαδικασία αύριο τελειώνει. Σας το θυμίζω, θυμίστε και στους συναδέλφους από κάθε πολιτική ομάδα. Αύριο στις 10 το πρωί έχουμε εκτακτή συνεδρίαση απλώς για να ψηφίσουμε. Να έχετε λοιπόν τις κάρτες σας μαζί. Στο, το 200 στο Winston Churchill θα γίνει η ψηφοφορία. Περίπου μια ώρα γιατί έχουμε διάφορες ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.